Καλημέρα σας ε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση και θα προχωρήσουμε αμέσως στο εργαστήριό μας για τις νέες άμεσες ενισχύσεις και τη νέα κατανομή στη μελλοντική κοινή αγροτική πολιτική και... ασχοληθεί με ένα από τα πιο δύσκολα και πιο λεπτά προβλήματα της μεταρρύθμισης, το νέο καθεστώς των άμεσων πληρωμών. Σκοπός είναι η αναδιανομή στα πλαίσια της μελλοντική ΚΑΠΑ. Καλωσορίζω τον Άλαν Σουίνμπαρκ που θα μας παρουσιάσει τις απόψεις του για το θέμα αυτό. Και μετά, ο συνήθως, θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση και ο καθηγητής θα απαντήσει στις ερωτήσεις και στα σχόλια των συναδέλφων. Καλωσορίζω και τον κύριο Μπότσορ και Κοντούρνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο κύριο Σουίνμπανκ από το Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ. Έχει το λόγο. Είπε ένα uh, Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Χαίρομαι που με καλέσατε να μιλήσω στην Επιτροπή σας σήμερα το απόγευμα Έχω μία παρουσίαση ε, PowerPoint. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες ε, διαφάνειες με γραφικές παραστάσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσετε να τις δείτε καλά. Αυτό που μου ζήτησα να κάνω, προετοιμάζοντας το σημείωμα που είδατε ορισμένοι από εσά, είναι να πάρω την πρόταση της Κομισιόν για τις άμεσες ε, πληρωμές, το νέο καθεστώς ε, άμεσων πληρωμών και να το αναλύσω με κριτικό βλέμμα. Δεν ήρθα εδώ λοιπόν σήμερα το απόγευμα για να σας πω τι πάει στραβά με την ΚΑΠ ή τι πρέπει να κάνετε με την ΚΑΠ. Ε, το καθήκον μου είναι πολύ πιο περιορισμένο. Θα μιλήσω δηλαδή για τις σημερινές προτάσεις που αφορούν τις άμεσες πληρωμές. Είναι ήδη επιτάπητος, το ξέρετε, και αρχίζουν να επηρεάζουν σίγουρα τη συζήτηση. Αξίζει να πούμε ότι πιστεύω ότι... Μάλιστα, επειδή υπάρχει και ένα δεύτερο σημείωμα για το, το στοιχείο του πρασινίσματος των άμεσων πληρωμών, τα σχόλιά μου δεν θα εστιάσουν πολύ στο πρασίνισμα, παρότι θα κάνω και κάποιες ε, παρατηρήσεις εκεί, ε, δεδομένης της σημασίας τους που έχουν στον ΠΟΕ. Επομένως, η παρουσίασή μου παρακολουθεί λίγο τη μορφή που έχει η έκθεση, έχει κάποια αρχικά σχόλια για τις ε, άμεσες πληρωμές ε, και τις επιπτώσεις τους πριν μπούμε στην ουσιαστική συζήτηση. Θέλω να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι το σύστημα των άμεσων πληρωμών που έχουμε στην ΚΑΠ ε, δημιουργήθηκε με έναν τρόπο ad hoc. Ξεκίνησε από την μεταρρύθμιση Μαξάρων πριν από 20 χρόνια μεταξελίχθηκε με τα χρόνια και σύν το χρόνο η έννοια των άμεσων πληρωμών άλλαξε από αντιστάθμιση που ήταν αρχικά σε στήριξη εισοδήματο των γεωργών. Ε, οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα προσπάθησαν να κρατήσουν τα ωφέλη των αγροτών, δηλαδή η μεταρρύθμιση Μαξάρων στήριζε τους γεωργούς για την απώλεια εισοδήματος ε, λόγω των ε, μειώσεων των τιμών στο Βόλιο και στα Δημητριακά και το 2003 με τη μεταρρύθμιση συνεχίσαμε. Ε, επιτρέψαμε στους γεωργούς να λαμβάνουν τις άμεσες πληρωμές που είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν, χωρίς όμως υποχρέωση να παράγουν γεωργικά προϊόντα. Η αποσύνδεση λοιπόν των άμεσων ενισχύσεων είναι πολύ βασικό τμήμα της κοινή γεωργικής πολιτικής και αποτελούν το 70% του προϋπολογισμού της ΚΑΠ το 2012. Είναι πολύ σημαντικό τμήμα λοιπόν αυτού. Θα ήθελα τώρα να σταθούμε μία στιγμή στις πιθανές επιπτώσεις των άμεσων πληρωμών. Με ανησυχεί το ότι οι άμεσες ε, πληρωμές είναι ένας ε, μηχανισμός που μπορεί να μην λειτουργήσει. Δεν πιστεύω ότι θα διαρκέσει η επίπτωσή του στο εισόδημα των ε, αγροτών. Γιατί υπάρχει μια αλληλεπίδραση και πιστεύω ότι άμεσες πληρωμές ουσιαστικά θα σημαίνει υψηλότερο κόστος, υψηλότερο κόστος για τη γη. Φυσικά οι δικαιούχοι θα αποφεληθούν αρχικά, αλλά θα ζημιωθεί συνολικά ε, χρόνο ο γεωργικός τομέας. Καθώς θα περνάει ο χρόνος, αν βλέπετε τους ε, λογαριασμού για τη γεωργία, ε, θα δείτε ότι η γεωργία ε, θα εξαρτάται πάρα πολύ από τις άμεσες πληρωμές. Είναι γενές στοιχείο τους. στοιχείο. Και ιδίω για τους νέους γεωργούς που θέλουν να αγοράσουν, να νοικιάσουν γη, ο πολιτής της γης θα γνωρίζει πάρα πολύ καλά το σύστημα των άμεσων πληρωμών και το ότι θα μπορεί να προσελκύσει αυτός ο νέος ας πούμε, γεωργός και αυτό θα ενσωματωθεί στο κόστος. Το, νέο, το πρόβλημα λοιπόν που αντιμετωπίζουν όσοι θέλουν να μπουν στο επάγγελμα είναι το, νέο, το υψηλό αρχικό κόστος. Ε, επομένως θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα των, αρχικών, των άμεσων πληρωμών. Ε, ανάγκασαν, καταδίκασαν δηλαδή τους γεωργούς ε, σε αυτές τις πληρωμές ε, που όλο και φουσκώνουν λόγω του ότι υπήρχαν στο παρελθόν και δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Ε, για ποιο λόγο υπάρχουν οι άμεσες πληρωμές. Η Κομισιόν έχει εκπονήσει πολλά έγγραφα για να στηρίξει τις σημερινές της προτάσεις. Ομολογώ ότι δεν μπορώ να βρω μια σαφή δήλωση για το τι, για ποιο λόγο υπάρχουν οι άμεσες πληρωμές. Η πιο σαφής δήλωση είναι ότι οι άμεσες ε, αποσυνδεδεμένες πληρωμές δίνουν βασικό, βασική στήριξη στο εισόδημα και στήριξη για τα βασικά δημόσια αγαθά που επιθυμεί η ευρωπαϊκή κοινωνία. Αν ανατάξετε στις συνθήκες, στη συνθήκη μάλλον. Υπάρχει ένα στόχος, να εξασφαλίσουμε δίκαιο επίπεδο ε, διαβίωσης για τους γεωργούς, αυξάνοντας ε, τα έσοδα των ατόμων που ασχολούνται με τη γεωργία. Το οποίο απεικονίζει το πώς εξελίχθηκε, πώς διαμορφώθηκε η γεωργική πολιτική. Με τη λέξη φέα, με τη λέξη δίκαιο, ε, ως οικονομολόγος, ε, έχω κάποιο πρόβλημα. Ε, η δικαιοσύνη είναι μια λέξη που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί. Ο καθένα έχει την άποψή του για τη δικαιοσύνη. Μιλάει για δίκαιο επίπεδο διαβίωσης της ε, γεωργικής κοινότητας. Ποια είναι, αυτή η γεωργική κοινότητα. Ας πούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι που παίρνουν ιστό. Ε, για αυτούς μιλάμε, για τους γεωκτήμονες μιλάμε. Για ποιους μιλάμε. Ε, ούτε αυτοί που φτιάχνουν την πολιτική γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί. Και μιλάει για την αύξηση των εσόδων των ατόμων που ασχολούνται με τη γεωργία. Αυτή η διατύπωση. Αυτός είναι ο στόχος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάτω επανάληψη δήλωσαν ότι τα εισοδήματα των γεωργών είναι χαμηλότερα από τα υπόλοιπα των υπόλοιπων εργαζομένων και σε ένα ψήφισμα του, του Ιουνίου του 2011 ε, αναφέρεται ότι τα εισοδήματα αυτά είναι ουσιαστικά χαμηλότερα κατά 40% από το, τα υπόλοιπα, τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας. Και το συμπέσμα της Κομισιόν από αυτό είναι ότι αν αυτά τα εισοδήματα είναι χαμηλότερα από τα υπόλοιπα, τότε θα πρέπει να συνεχίσουμε να τα στηρίζουμε αυτά τα εισοδήματα. Μπορεί όμως να συνέχει κανείς άλλα συμπεράσματα. Είχαμε ούτως ή άλλως 20 χρόνια πίσω μας ε, άμεσων πληρωμών ε, και συνολικά 50 χρόνια στήριξης των γεωργικών εισοδημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν είναι καταγγελία, κατηγορία της αποτυχίας της ΚΑΠ αυτή, ότι στηρίζουμε τόσα χρόνια, 50 χρόνια ας πούμε, τα εισοδήματα αυτά, αν ισχύουν αυτά τα νούμερα τα έσοδα από την εμπορική γεωργία είναι πραγματικά χαμηλότερα από αυτά που πετυχαίνει κανείς από τους υπόλοιπου ε, οικονομικούς τομείς. Δεν νομίζω ότι έχουμε σαφή εικόνα. Αν πάω πάλι στην ε, αξιολόγηση επιπτώσεων της Κομισιόν, λέει ότι δεν έχουμε πολλά στοιχεία για τα εισοδήματα ε, των γεωργικών οικοκυριών. Άρα δεν σχολιάζει τι διάφορε επικρίσεις που έχουν ασκηθεί σε ό,τι αφορά την εμπορική πάντα γεωργία. Ε, δεν είναι κατά ανάγκη αληθές ότι τα εισοδήματα αυτά των ε, γεωργικών νοικοκυριών ε, είναι χαμηλότερα από τα υπόλοιπα. Όταν κοιτάς τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα άμεσων πληρωμών λειτουργεί, δεν υπάρχουν στοιχεία. Ε, δεν υπάρχει έλεγχος των εισοδημάτων. δεν υπάρχει έλεγχος του κατά πόσο αυτός που λαμβάνει αυτή τη στήριξη έχει την ανάγκη. Όσοι δεν έχετε μπροστά στη διαφάνεια, ίσω ίσως και στο βάθος δεν βλέπετε καλά. Πάντως, η, η κατανομή εισοδήματο στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2010, βλέπετε, ε, στην, ε, στις κόκκινες τους δικαιούχους και στις μπλε στήλε, τις δαπάνες. Αριστερά έχουμε στο άξονα των ε, ψη 0 μέχρι 35 ε, και στον άξονα των Χ έχουμε από 0 έως 500 ευρώ και φτάνουμε μέχρι πάνω από 500.000 ευρώ ε, δεξιά στον άξονα των Χ. Αν πάμε σε εισοδήματα κάτω από 500 ευρώ, έχουμε 44% των ε, δικαιούχων που, παίρνουν, που έχουν αυτά τα εισοδήματα και είναι το 4,2%. Ενώ πάνω από 500.000 ή μάλλον το 9% των χρημάτων ε, το παίρνουν άνθρωποι με εισοδήματα πάνω από 150.000 ευρώ. Προσπαθούμε να αναλύσουμε και να καταλάβουμε αυτά τα νούμερα. Υπάρχουν πολλές ε, περιπτώσεις εδώ, αλλά δεν υπάρχει λογική σύνδεση ανάμεσα σε αυτή την ανάγκη στήριξης των εισοδημάτων των διοργών και τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα. Η Κομισιόν μιλάει για δημόσια αγαθά επίση. Δεν είναι πάντα εύκολο να καταλάβουμε τι έχει στο μυαλό της η Κομισιόν όταν μιλάει για αυτή την έννοια. Από ό,τι φαίνεται στις προτάσεις της υπάρχουν τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι τα βασικά δημόσια αγαθά. Εδώ υπάρχει σχέση με την πολλαπλή συμμόρφωση και τις καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Γιατί είναι απαραίτητο, διερωτώ με, να πληρώσουμε τους γεωργούς για να τηρήσουν τον νόμο. Αν αυτά τα προβλέπει το γεωργικό σύστημα, γιατί να μην τα τηρήσουν. Σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο υπάρχουν πάντα κάποιες προϋποθέσεις και πρέπει να τις τηρούμε. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί πρέπει να πληρώσουμε, να αντισταθμίσουμε, να επιβραβεύσουμε τους ε, γεωργούς ε, γιατί τηρούν τον νόμο. Και η πολυλειτουργικότητα αφορά τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και τα λοιπά χαρακτηριστικά που η Γεωργία ε, εξασφαλίζει στην υπόλοιπη κοινότητα ε, και τα οποία α, τα θέλει η υπόλοιπη κοινότητα. Γιατί είναι, σε, είναι σπάνια αυτά τα, χαρακτηριστικά και θα πρέπει να τους ανταμείψουμε τους γεωργούς που μας τα δίνουν. Ε, με το σύστημα των άμεσων πληρωμών η εξασφάλιση της πολιτουργικότητας βασίζεται στον αλτρουισμό των γεωργών. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία συμβατική υποχρέωση να μας δώσουν μια πολυλειτουργική γεωργία. Το τρίτο στοιχείο το οποίο προκύπτει από, το από τα έγγραφα είναι ότι πληρώνουμε για την επιστηστική ασφάλεια. οι Ευρωπαίοι γεωργοί αντιμετωπίζουν ψηλότερο κόστο, το οποίο θα πρέπει να αντισταθμιστεί γιατί παράγουν, υποτίθεται, τροφή πιο ασφαλή από, την, από τα εισαγόμενα τρόφιμα. Αν τα εισαγόμενα τρόφιμα είναι λιγότερο ασφαλή, τότε κάτι να κάνουμε με τα εισαγόμενα ε, τρόφιμα. Όχι να κάνουμε κάτι αντίστροφα για τα δικά μας. Αν δεν είναι ε, ασφαλή αυτά τα τρόφιμα, τα εισαγόμενα, δεν θα πρέπει να πολλούνται στην αγορά, απλούστατα. Οι προτάσεις της Κομισιόν είναι ένα, μια δέσμη ε, δύσκολων, περίπλοκων προτάσεων. Δεν είχα το χώρο στην έκθεση και το χρόνο τώρα να διατρέξω όλα τα επιμέρους θέματα. Θέλω να σταθώ όμως ε, σε κάποια σημεία, τα οποία αυτά που βλέπετε εδώ στην διαφάνεια. Καταρχάς, ε, ο προπολογισμό για τις άμεσες πληρωμές. Η Κομισιόν έκανε τεράστια προσπάθεια για να εξασφαλίσει τον προπολογισμό της ΚΑΠ και την κατανομή της που θα παραμείνει ανέγκυχτη λίγο πολύ μέχρι το 2020. Αυτό ε, σημαίνει ουσιαστική μείωση καθώς θα αυξάνεται ο πληθωρισμός. Αλλά βασικά το παλιό σύστημα με κάποιες μικρές αλλαγές ε, συνεχίζεται δημοσιονομικός πώς ε, και περνάει στο νέο σύστημα. Αυτό είναι πολιτική απόφαση και ως οικονομολόγος τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα. Γιατί δεν γίνεται καμία προσπάθεια για να δικαιολογήσουν τον προπολογισμό των άμεσων πληρωμών με μια προσέγγιση που συγκεντρώνει ιδέες από κάτω ας πούμε, και τις στέλνει σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Όχι, είναι μια πολιτική απόφαση. Ε, δικαιολογείται ίσως πολιτικά, ε, γιατί θέλουν ε, να έχουν επιχείρημα στις διαπραγματεύσεις, αλλά νομίζω ότι η Κομισιόν και εσείς οι Ευρωβουλευτές χρειάζεστε και ένα σχέδιο σε περίπτωση που το πρώτο σχέδιο αυτό, το, το πρώτο σχέδιο δεν πάει καλά. Ένα plan B δηλαδή. Δεν θέλετε να πάτε σε διαπραγματεύσεις και να πείτε δεχόμαστε μια μείωση 20%. Αν, ας πούμε, οι Υπουργοί Οικονομικών αποφασίσουν τη μείωση κατά 20% της ΚΑΠ, αυτό σημαίνει 8 δισεκατομμύρια ε, ευρώ που είναι ε, λιγότερα, που είναι ε, το 80% του δεύτερου πυλώνα. Τι θα κάνετε τότε θα εξαλείψετε τον πυλώνα 2, τον δεύτερο πυλώνα και θα κρατήσετε τον πρώτο, πίνα, ε, τον πρώτο πυλώνα. Θα πρέπει να αποφασίσετε τι προτιμάτε, τι θέλετε. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις ε, για αναδιανομή μεταξύ των κρατών μελών με ένα περίπλοκο μαθηματικό τύπο. Ίσως όχι και τόσο περίπλοκο, αλλά τα κράτη-μέλη που το μέσο ποσοστό ε, αναεκτάριο μάλλον το μέσο ποσοστό νεκτάριο αυξάνεται και σε άλλα που μειώνεται. Ε, χρησιμοποιείται πολύ η λέξη δικαιοσύνη πάλι ε, στη, στην όλη συζήτηση. Το θέμα είναι, θα είναι αποδεκτό στις χώρες αυτές που έχουν ένα επίπεδο πληρωμής ε, κάτω από το μεσόωρο. Ε, θα είναι πολύ σκληρό για αυτές που είναι πάνω από το μεσόωρο και αν θα, υπάρξουν, θα υποστούν ε, μειώσεις. Δεν υπάρχει απάντηση, ας πούμε, τεχνική, είναι πολιτική απόφαση. Γιατί στην ε, τεκμηρίωση ε, δεν γίνεται καμία απόπειρα για να δικαιολογηθούν οι άμεσες πληρωμές. Δεν αναφέρεται η στήριξη του εισοδήματος στα δημόσια αγαθά, η συνοχή, ότι προσπαθούμε να δώσουμε λεφτά σε φτωχότερες ε, περιοχές της υπαίθρου για να καθορίσουμε την ανακατανομή. Όχι βλέπετε τι, έχουμε, τι είχαμε στο παρελθόν, θα τα κάνουμε έτσι μια, ένα χτένισμα, έτσι μια, ένα μασάζ αν θέλετε, ε, για, να τα, για να τα καταπιούν καλύτερα ας πούμε. Δεν υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα που να καθορίζει ποιε πρέπει να είναι αυτέ οι άμεσε πληρωμέ. Ούτω ή άλλω. Για το πρασίνισμα τώρα, Πρόεδρε. Η πρόταση τη Κομισιόν λέει ότι το 30% των ποσών που πηγαίνει σε ένα κράτο μέλο θα πρέπει να μπει σε, αυτό σε αυτή τη συνιστόσα του πρασινίσματο, σε αυτό το κουτί του, πρασινίσματο, του πρασινίσματος, το κείμενο τη Κομισιόν με μπέρδεψε. Καταρχά αφελώ υπέθεσα ότι υπήρχαν δύο πληρωμέ. η βασική πληρωμή και η πράσινη πληρωμή. Αλλά αν διαβάσετε το κείμενο πιο προσεκτικά, ε, φαίνεται ότι είναι μία η πληρωμή τελικά, που έχει απλώ δύο συνιστώσει. τη βασική πληρωμή συν την πράσινη πληρωμή. Και δεν είναι διχωριστέ αυτέ τι πληρωμέ, είναι απλώ δύο συνιστώσει τη ίδια ε, πληρωμή. Και αυτό είναι πολύ επιτακτικό. Ε, αν, α πούμε, είσαι μια κλασικό γεωργό σε αεροτρέα καλλιέργεια, α πούμε, θα πρέπει να έχει τρει σοδιέ. Επίση, ε, δεν υπάρχει κατανομία εθνική, σε εθνική βάση ή περιφερειακή βάση, δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια. Φυσικά υπάρχουν οι δηλώσει για τα περιβαλλοντικά ωφέλη, ναι, αυτό το δέχομαι. Αλλά είναι δύσκολο να συνδέσουμε τις πραγματικές πληρωμές που θα πάρει ένας γεωργός ή τις πληρωμές που θα πάρει ένας γεωργός σε μια περιοχή με τα περιβαλλοντικά ωφέλη, ας πούμε, που θα προκύψουν. Το κόστος με βάση την Κομισιόν και τη μελέτη αντικτύπου της θα είναι 33 ε, με 41 ευρώ ανεκτάριο που για μερικούς θα είναι μεγάλο το κόστος, αλλά θα Και η μέση πληρωμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι 80 ευρώ το εκτάριο. Φυσικά σε μερικές χώρες θα είναι υψηλότερο ή χαμηλότερο από αυτό. Εξαρτάται από το αν αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάνω ή κάτω από το μέσο όρο ό,τι αφορά τις άμεσες πληρωμές. Όλα αυτά τα θέματα, και θα επανέλθω σε αυτά σύντομα, ε, δημιουργούν μείζωνα προβλήματα ε, στον ΠΟΕ. Ή θα δημιουργήσουν μείζωνα προβλήματα στον ΠΟΕ. Η ενεργή γεωργή. Και πάλι. Δικαιοσύνη, διαφάνεια, ε, πιο αποδεκτή πολιτική από το κοινό. Ε, υπάρχουν επικρίσεις όμως από το Ελεκτικό Συνέδριο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι αυτοί είναι λόγοι για να κάνουν την Κομισιόν να υποβάλει αυτή την πρόταση, υποτίθεται. Τώρα ως οικονομολόγος δεν βλέπω γιατί πρέπει να πιστέψουμε ότι η ιδιοκτησία των εκμεταλλεύσεων, η διαχείριση των εκμεταλλεύσεων αυτών θα επηρεάσει ή το να είσαι μάλλον θα επηρεάσει την διαχείριση της γης. Επίσης, φεύγουν κάποιες γης από την πολλαπλή συμμόρφωση. Αυτό είναι θετικό, υποτιθέται. Εγώ δεν είμαι γεωργός, πρόεδρε. Όταν ήμουν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο όμως, το πανεπιστήμιό μου ε, διαχειριζόταν ε, μία μεγάλη εμπορική α, γεωργική εκμετάλλευση με αεροτρές καλλιέργειες. Και παρήγαμε μία πολυλειτουργική γεωργία. Διαβάζοντας την πρόταση της Κομισιόν, Επειδή οι άμεσες πληρωμές ε, αυτών των γεωργών είναι λιγότερες από το 5% των εισοδημάτων του Πανεπιστημίου, ε, δεν θεωρείται, ουσιαστικά εξαιρούνται αυτοί οι γεωργοί από το σύστημα. Can be ε, so that it... Πώς λοιπόν θα αποφύγουμε ότι υπάρχει υποχρέωση παραγωγής να είναι κάποιος δηλαδή ενεργός, εν ενεργεία αγρότης. Πώς θα βρούμε ένα σχήμα που δεν θα παραβιάζει τους κανόνες του ΠΟΕ. Υπάρχουν ε, πολλές προτάσεις για τα νότατα όρια, για τους μικρούς ε, αγρότες, ε, τους νέους και τη μερική σύζευξη ή σύνδεση και όλα έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση κάποιων πολιτικών μελημάτων. Φαντάζομαι ότι εσεί είστε στην καλύτερη θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να λάβετε τι αποφάσει. Εγώ πολύ λίγα μπορώ να πω πάνω σε αυτό, αλλά πρέπει να σα πω ότι για καμία από αυτέ τι προτάσει δεν βρίσκω κάποια οικονομική λογική, γιατί νομίζω ότι οι δυνάμει μπορούσαν όλε να ε, παρεμποδίσουν τελικά τι απαιτούμενε δομικέ αλλαγέ που πρέπει να επιτελεστούν αν θέλουμε η γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ανταγωνιστική. Όσο δε ε, για τους ε, ερχόμενους υπάρχουν ε, και τα αντίθετα αποτελέσματα. Με αποτέλεσμα η πρόταση αντί να αντιμετωπίζει το πρόβλημα, αντιμετωπίζει το σύμπτωμα. Πάλι ε, σας δείχνω ένα γράφημα, δεν ξέρω αν θα το δείτε όλοι. Αυτό που βλέπετε όμως, όσοι βλέπετε, είναι η ετήσια δήλωση ε, της ε, εγχώριας στήριξης που αποστέλει κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση στον ΠΟΕ. Ξεκινάμε από το έτος 95-96 και καταλήγουμε πριν από 10 μέρες τουλάχιστον το έλεξα, κατέληξαμε στο έτος 2007-2008 σε αυτή τη χρήση. Κάτω-κάτω έχουμε το λεγόμενο και χρυμπάνιο κουτί Amber Box, ε, τα πορτοκαλιά, η πορτοκαλιά στήλη. Εκεί υπάρχουν κάποια όρια. Από πάνω έχουμε το μπλε κουτί που δεν σταυρώνει τόσο πολύ το εμπόριο και το green box από πάνω, οι πράσινε στήλε, το πράσινο κουτί. Οι πολιτικέ μεταρρυθμίσει ουσιαστικά από το κεχριμπαρί το πήγαν, πήγαν στο μπλε ε, κουτί τη στήριξη ουσιαστικά και από το 2003, τις μεταρρυθμίσεις του 3 και μετά, από το πορτοκαλί ή και χρυμπαρί και το μπλε, η στήριξη πήγε στο πράσινο κουτί. Βλέπουμε λοιπόν ε, την, ε, τα ποσά, ε, είναι τα όρια ουσιαστικά αυτή η γραμμή που βλέπετε και υπολείπεται πάρα πολύ η, η στήριξη σε ό,τι αφορά την σύνδεση. Δεν έχουν, δεν έχουν δηλαδή εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους ό,τι αφορά το EMS binding δηλαδή την ε, ομαδοποιημένη μέτρηση της στήριξης, AMS, 72,2 δισεκατομμύρια είναι το ποσό. Εάν έχουμε έκβαση στο γύρο της Ντόχας, καταλαβαίνω ε, ή θα καταλάβω αν κάποιοι μη διάσετε μέσα στην αίθουσα, ε, ακούγοντας αυτό που λέω για το γιο. αλλά τέλος πάντων έχουμε μία πρόταση για μείωση του AMS Binding κατά 70%. Αν επιβληθεί κάτι τέτοιο, τότε για την Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσό το αντίστοιχο θα είναι 21,7 δισεκατομμύρια. Όπως είπα στην πράξη, η δήλωση για το έτος 2007-2008 ήταν πάρα πολύ χαμηλή, μόνο 12,4 δισεκατομμύρια. Δηλαδή και είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω, ε, υπολείπεται του επίπεδου των υποχρεώσεων, των δεσμεύσεων, αλλά μάλλον θα είναι ε, και χαμηλότερη σε σχέση και με τις ε, δεσμεύσεις που ενδέχεται να αναλυφθούν στο πλαίσιο του γύρου της Ντόχας. Επίσης έχουμε το ε, σχήμα των ε, άμεσων πληρωμών SPS και SAPS για το 2007-2008. Τα ποσά ανέρχονταν σε 34,5 δις. Εάν αυτό το σχήμα των ε, άμεσων πληρώμων, το SPS και το διάδοχο σχήμα με βάση την πρόταση της Κομισιόν δεν είναι μέτρα πράσινου κουτιού, και αν προσθέσουμε αυτά τα 34,5 δις ε, ε, στα 12,4 δις στο AMS, εκεί δημιουργούμε προβλήματα. Πώς μπορούν λοιπόν να μπέσουν στο, στα μέτρα πράσινου κουτιού τελικά ε, αυτά τα μέτρα. Θα πρέπει οι δηλώσεις αυτές τελικά να γίνονται από τον ΠΟΕ. Δηλαδή δεν κάθεται ο γραμματέας του ΠΟΕ και βάζει στα τετραγωνίδια, δεν τσεκάρει τα τετραγωνίδια απλά για να πει ναι καλά ή όχι. Σε κάποια φάση στο τέλος ε, ίσως ε, ε, χρειαστεί να υπάρξει να κινηθεί ο μηχανισμός ε, της επίλυσης διαφορών. Οπότε εκεί πηγαίνουμε σε απαιτήσει πράσινου κουτιού. Μία θεμελιώδη απέτηση του πράσινου κουτιού, των πολιτικών πράσινου κουτιού, είναι να είναι ως το δυνατόν λιγότερο ή μηδαμινό, ε, μηδενικό το στρεβλωτικό τους αποτέλεσμα. Ή η Ευρωπαϊκή Θεσμή, Θεσμικά Όργανα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λοιπόν το λέω αυτό, έκανε κάποιες δηλώσεις ε, που... Πού είναι αυτές οι πολιτικές που δεν έχουν καμία επίπτωση. Παραδείγματος χάρη τον Ιούλιο του 2010 δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, μια βασική άμεση χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους ε, Ευρωπαίους, τους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξασφαλιστεί η οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού μοντέλου γεωργικής παραγωγής για να υπάρχει βασική επιστηστική ασφάλεια. Δεν ξέρω τι εννοείται ακριβώς με αυτό τον όρο, φαντάζομαι εννοείται περισσότερα τρόφιμα να παράγονται στην Ευρώπη. Επίσης λέει ότι θα πρέπει να μπορούν οι αγρότες να παράγουν ανταγωνιστικά ε, ποιοτικά τρόφιμα. Δεν καταλαβαίνω τι θα πει αυτό. Το ανταγωνιστικά και επίσης λέει ότι θα πρέπει η δραστηριότητα και οι θέσει εργασία στις ε, περιοχές υπαίθρου να ενθαρρυνθούν κτλ. Μήπως η βραζιλιανή κυβέρνηση στο μέλλον ε, χρειαστεί αυτή τη δήλωση στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Καλό είναι να το καταγράψει. Λέτε εδώ ότι πρέπει να παραμείνει η γεωργική παραγωγή στην Ευρώπη. Αλλά αυτό δεν τηρεί τις βασικές απαιτήσεις του πράσινου κουτιού. Και μετά υπάρχουν και κάποια ειδικά κριτήρια πολιτικής. Παραδείγματο χάρη, εάν θέλει κανείς ε, να δηλώσει πληρωμές ως αποσυνδεδεμένη στήριξη εισοδήματο, τότε με βάση την υποπαράγραφο 6 Δέλτα, οι πληρωμές αυτές δεν θα πρέπει να σχετίζονται να βασίζονται στους παράγοντες παραγωγής που εφαρμόζονται οποιοδήποτε έτος μετά το έτος βάσης, την περίοδο βάσης. Δηλαδή το δικαίωμα δεν εγγυάται ότι θα έχει την πληρωμή. Θα πρέπει το δικαίωμα να ενεργοποιείται σε αιτήσια βάση και να περιλαμβάνει και τις επιλέξιμες γεωργικές γέες που υπόκεινται στην ε, πολλαπλή συμμόρφωση μεταξύ άλλων και το GAEC. Μα τελικά μπορεί κάποιος να πει συνδέεται τις πληρωμές με παράγοντες παραγωγής. Production factors. Ερχόμαστε τώρα ε, σε ακόμα πιο προβληματικά θέματα όπως αυτά των ενεργεία αγροτών και του πρασινίσματος. Ε, στο 6ε λέγεται ότι δεν απαιτείται παραγωγή για την ε, λήψη πληρωμής. Επομένως, τι λέει ουσιαστικά, τι θέλει το ΟΠΟΕ, μη ενεργούς, ανενεργούς αγρότες. Και αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι ενεργεία αγρότες παράγουν κάτι, τελικά ε, πάρα πολύ δύσκολο μπορεί κανείς να το περάσει αυτό με στον ΠΟΕ. Να πείσει ένα πάνελ, μια επιτροπή, ότι δεν απαιτείται παραγωγή για, την, ε, για να μπορεί κανείς να λάβει τις πληρωμές. Και επανέρχομαι στο πρασίνισμα. Πρέπει να παρέχει κανείς τρεις καλλιέργειες. Και δεν καταλαβαίνω εγώ αυτή η απέτηση περί πρασινίσματος πώς μπορεί να εγγραφεί χωρίς αυτό να σημαίνει απέτηση για παραγωγή. Εάν τώρα το πρασίνισμα αφορά μία πληρωμή και αν αυτές είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και δεν είναι δύο οι πληρωμές, τότε συνολικά, συνολικά η βασική πληρωμή δεν μπορεί να μπει στο πράσινο κουτί. Αν μπορούμε βέβαια να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο, το πρασίνισμα δηλαδή από τη βασική συνιστόσα, τότε έχουμε μεγαλύτερο ε, έδαφος μπροστά μας να κινηθούμε. Πού θα μπορούσε λοιπόν να πάει αυτή η συνιστόσα πρασινίσματος. Γίνεται λόγος για την επιλεξιμότητα των πλέον στην παράγραφο 12 και λέω ότι πρέπει να καθορίζονται η επιλεξιμότητα στο ως πλαίσιο ενός πολύ σαφώς καθορισμένου κρατικού περιβαλλοντικού προγράμματος προγράμματος συντήρησης και ότι θα πρέπει εξαρτάται από την εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων στο πλαίσιο του κρατικού προγράμματος περιλαμβανομένων ε, των όρων που σχετίζονται με τις μεθόδους παραγωγής ή τα input και μετά λέει ότι το ποσό της πληρωμής περιορίζεται στο επιπλέον κόστος ή απώλεια εισοδήματος που ε, συνεπάγεται από την ε, συμμόρφωση προς αυτό το κρατικό πρόγραμμα. Άρα διπλάσιο τριπλάσιο θα είναι το ποσό της πληρωμής από το κόστος συμμόρφωσης προς το πρόγραμμα. Αν καταλαβαίνω καλά αυτά που διαβάζω στο έγγραφο της Κομισιόν. Έτσι ε, έχουν τώρα τα πράγματα και αυτό έχει κάποια σημασία. Αυτή τη στιγμή όχι γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ μεγάλο πεδίο, πολύ σχόρος ακόμα ε, στο και χρυμπαρί και μπλε κουτί. Αλλά είναι και απίθανο ότι θα ασχοληθεί κάποιο μέλος του ΠΟΕ για να ε, προκαλέσει να προσβάλλει όλη αυτή τη διαδικασία. Εάν τώρα το πακέτο της Ντόχας εγκριθεί δύσκολα, μπορεί. Τώρα Πού, μέχρι πού μπορούμε να φανταστούμε ε, στο μέλλον τι θα πάμε με όλους αυτούς τους αστάθμιτους παράγοντες. Δεν ξέρω. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έχω μακρηγορήσει πάρα πολύ, γι' αυτό έρχομαι σε κάποιες συστάσεις. Ίσως να μην θέλετε να βάλετε στο χαρτί ε, με μελάνι το εναλλακτικό σας σχέδιο. Σκεφτείτε το τουλάχιστον όμως. Μήπως θα έπρεπε για τις μειώσεις να στοχεύσετε στον πυλώνα 1 και όχι στο 2. Είναι μια πρόταση. Και αντί να έχετε το πρασίνισμα στον πρώτο πυλώνα θα μπορούσατε αυτό το 30% των ε, κονδυλίων να τα ε, μεταφέρετε στον πυλόν 2 που μπορεί να συνδέονται με την παράδοση των αποτελεσμάτων ε, οι πόροι και θα μπορούν τα κράτη-μέλη να σχεδιάζουν προγράμματα πιο καλά προσαρμοσμένα στις ε, συνθήκες εκάστοτε ή ίσως ε, να εξασφαλίσετε ότι η συνιστόσα του πρασινίσματος είναι εντελώ ξεχωριστή από τη βασική πληρωμή. Οπότε έτσι θα έχουν τα κράτη-μέλη πολύ μεγαλύτερη δεκριτική ευχαίρεια για να καθορίσουν τους κανόνες για τη συνιστόσα αυτή του πρασινίσματος. Επίσης, μήπως θα έπρεπε να εγκαταληφθούν οι προτάσεις για τους ενενεργοί αγρότε. Να αποφευχθεί οποιαδήποτε υπόδειξη ή ε, υπόθεση ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει σχέση ε, άμεσων πληρωμών με τη διαθεσιμότητα τροφίμων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πρόκειται για αποσυνδεδεμένε πληρωμές. Φοβούμε ότι δεν είναι η τελευταία αυτή, η τελευταία μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική. Νομίζω ότι μετά από πέντε χρόνια θα εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα με τη Γεωργία. Οι φορολογούμενοι θα εξακολουθούν να διερωτώνται αν τα χρήματά του δαπανώνται με το σωστό τρόπο και οι κυβερνήσει θα εξακολουθούν να πιστεύουν ότι στρεβλώνεται ο ανταγωνισμό με το σύστημα των άμεσων πληρωμών. Μπορεί να μην είναι για την παρούσα, ε, αλλά αρχίστε να σκέφτεστε και το μέλλον, τη μελλοντική μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ. Και σα θέτω δύο ερωτήματα που μπορούν να σα απασχολήσουν. Αν στόχο ήταν η στήριξη τη ΚΑΠ, η στήριξη του εισοδήματο των αγροτών, τα τελευταία 50 χρόνια, γιατί εξακολουθεί να υφίσταται πρόβλημα με τα εισοδήματα των αγροτών. Και δεύτερο ερώτημα, τελικά ε, η ΚΑΠ, τι στόχο έχει. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Νομίζω ότι η παρέμβασή σας έχει ε, προκαλέσει ή μάλλον θα προκαλέσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση της οποίας το εναρκτήριο λάκτισμα θα δώσει ευθύ αμέσως. Κανιέτη πρώτα και μετά ο κύριος Ντόρφμαν. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τον προσκεκλημένο ομιλητή για την ενδιαφέρουσα και πλήρη παρουσίαση του θέματος που περιέχει και πολλά αναλυτικά συμπεράσματα. Ας μην λησμονούμε ωστόσο και την κλίμακα των διαφορών στις διάφορες, στους διάφορους τόπους παραγωγής ε, για την γεωργία. Συμφωνώ σε ορισμένα σημεία βέβαια στο κεντρικό θέμα που έχει σχέση με τις άμεσες ενισχύσεις. Η μεταρρύθμιση πάντως της ΚΑΠ θα πρέπει να διασφαλίσει δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των γεωργών και ταυτόχρονα δημιουργία θέσεων απασχολήσεως. Το σύστημα άμεσων ενισχύσεων στην ουσία θα καταστήσει ανάπηρη την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Γι' αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να συζητήσουμε περί κατοφλίων και περί οροφών όταν μιλούμε για τις άμεσες ενισχύσεις, για τον όγκο δηλαδή των άμεσων ενισχύσεων. Ορισμένοι παίρνουν πάρα πολύ λίγα και άλλοι παίρνουν υπερβολικά πολλά και είναι δύσκολο να εξηγηθεί γιατί κάθε φορά. Για το πρασίνισμα σε χώρες όπως η Λετωνία για παράδειγμα, όπου οι περισσότερες εκμεταλλεύσεις μας είναι μικρές, Ε, τα μέτρα αυτά θα είναι καταστροφικά. Και ιδιαίτερα για τη δασοκομεία. Θα πρέπει λοιπόν οι άμεσες νησίες να κατευθυνθούν εκεί όπου είναι απαραίτητε. Ρωτώ τώρα και τον κύριο καθηγητή αλλά και τον εισηγητή. Οι επικρίσεις κατά του καθεστώτος των άμεσων ενισχύσεων πράγματι δεν έχουν οικονομικό θεμελ, οικονομική θεμελίωση. Η ιδέα είναι περισσότερο να αντιληφθούν κονδύλια από τον πρώτο πυλώνα γιατί όπως είπε ο Επίτροπος θέλουμε να καταλήξουμε σε μια κατάσταση που να μην υπάρχουν ούτε πολύ χαμένοι ούτε πολύ κερδισμένοι. Οι άμεσες ενισχύσεις θα πρέπει να δίνονται με αντικειμενικά κριτήρια. αναλόγως και με το μέγεθος της, των, των γεών που θα μπουν στην παραγωγή και πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τις, τα πορίσματα των επιστημονικών ερευνών και βέβαια να εγκύψουμε στα θέματα που μας έχει αναθέσει η κοινωνία. Ευχαριστώ και τον κύριο καθηγητή για την διάλεξή του που μου φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αλλά και αρκετά προβοκατόρικη των εισαγωγικών για να μας ξυπνήσει ε, ένα τέτοιο απόγευμα, κάτι που δεν είναι και εύκολο. Θα αρχίσω με τα συμπεράσματά σας από το τέλος όπου έχετε δίκιο, δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε ήδη από τώρα τι θα κάνουμε σε 5-6 χρόνια σε ό,τι αφορά την ε, αναθεώρηση της ΚΑΠ. Τώρα, εάν το συνδέσω αυτό με την κάπως προβοκατόρικη πρότασή σας, γιατί δεν παίρνουμε ένα μέρος των κονδυλίων από τον πρώτο πυλώνα για να τον διαθέσουμε στον δεύτερο πυλώνα και να οργανώσουμε και καλύτερα, πιο λογικά περιβαλλοντικά προγράμματα και όχι αυτές τις ανοησίες του πρασινίσματος που προτείνονται τώρα για τον πρώτο πυλώνα, Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό πράγματι θα ήμασταν στη σωστή οδό. Δηλαδή βέβαια σε 5-6 χρόνια θα έχουμε ξανά το ίδιο ερώτημα. Πώς θα αιτιολογήσουμε τις πληρωμές του πρώτου πυλώνα. Και τότε θα πρέπει βέβαια να επινοήσουμε κάτι το νέο. Όπως έγινε την προηγούμενη φορά η λεγόμενη cross compliance, η πολλαπλή συμμόρφωση, τώρα το πρασίνισμα, τότε θα χρειαστεί να επινοήσουμε κάτι άλλο. Και δεν ξεφεύγουμε από τον ε, φαύλο αυτό κύκλο. Χρειάζεται λοιπόν σοβαρότερη αντιμετώπιση και πολύ πιθανό να έπρεπε να βασιστούμε περισσότερο στο δεύτερο πυλώνα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν είπατε ωστόσο τίποτε για το δικό μου αγαπημένο θέμα που είναι η κατανομή μέσα στις χώρες μέλη. Εγώ αναγκάζομαι εδώ τώρα να αναφέρω αριθμούς. Για παράδειγμα, στην πατρίδα μου, κατά μέσον όρο είναι 550 ευρώ το εκτάριο στην περιοχή, την πιο ευνοημένη περιοχή και αν εξετάσω τις εκμεταλλεύσεις οι οποίες στις αρχές της χιλιετίας μόλις δηλαδή υπολογίστηκαν οι αποσυνδεμένες, τα αποσυνδεμένα ποσά και έκαναν εκτροφή βοηδών, αυτές οι εκμεταλλεύσεις λαμβάνουν μέχρι και 1000 ευρώ ανά εκτάριο. για καλαμπόκι 719 ευρώ, άλλοι που είχαν άλλες καλλιέργειες λαμβάνουν 400 ευρώ ανά και ανεξαρτήτως του τι πράττει σήμερα. Ε, συγγνώμη, όχι αραβός αλλά ρύζι. Και υπάρχουν και οι ταλέποροι, οι οποίοι στην δική μου για παράδειγμα εκλογική περιφέρεια δεν λαμβάνουν παραπάνω 55 ευρώ το εκτάριο. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Μέσα στι ίδιε τι χώρες μέλη έχουμε προφανέστατε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και προφανέστατε ανισότητες, οι οποίες κατά τη γνώμη μου και πρέπει να συζητηθούν και πρέπει να απαλληφθούν. Η δεμή, η πορεία οδηγεί κατευθείαν στον γκρεμό. Δεν μπορεί να αιτιολογηθεί πλέον η ε, κατάσταση αυτή και βέβαια και οι αγρότησες και οι αγρότες δεν είναι πλέον διατεθειμένοι να ανεχθούν τις ανισότητες αυτές. Ότως ή άλλως μεταξύ χωρών μελών, ακόμη περισσότερο μεταξύ, μέσα στις ίδιες τις χώρες. Πρέπει να βρεθεί κάποια λύση λοιπόν. Να πούμε ίσως ότι κάθε περιφέρεια θα πρέπει να έχει περιφερειακή κατανομή των ε, κοντιλίων. Τότε ίσως να λυθεί βέβαια το πρόβλημα εντός των περιφερειών, δεν θα λυθεί όμως μεταξύ των περιφερειών. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι ευφυείς λύσεις που να προταθούν και να υλοποιηθούν από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο Γιάννοφ και μετά Άγνιο. <laughs> Um, Ωραία ήταν αυτή η... Μα δεν με κοιτάτε. Ε, ε, σας κάνω φιλοφρόνηση. <clears throat> Ήταν εξαιρετική έκθεσή σας και πραγματικά προκαλεί σκέψεις και πολύ καλά κάνατε και την κάνατε. Κάθε μορφή στήριξης καταλήγει στους λάθος ανθρώπους. Στη Βρετανία καταλήγει στους μεγάλους ε, κτηματίες. Και εγώ έχω, ε, αν και εγώ είμαι, ε, και εγώ είμαι κτηματίας και μου πούν θα πάρεις άμεσε ε, πληρωμές, βεβαίως. Αλλά αν είμαι αγρότης δεν βρίσκω μεγάλη ωφέλεια. Το ίδιο πρόβλημα θα υπάρχει για κάθε άλλη μέθοδο στήριξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η μοναδική που στηρίζει τη Γεωργία. Έχετε και τι Ηνωμένε Πολιτείε και τον Καναδά και την Ιαπωνία με, τα, με τον βασικό του νόμο. Όλοι αυτοί στηρίζουν τη Γεωργία. Αυτό δεν το είπατε βέβαια. Και ίσω θα έπρεπε να το κάνετε ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλο που την αντιπαθώ δεν είναι και η μοναδική στον κόσμο που κάνει τα πράγματα αυτά. Εκεί όπω όπου είμαστε μοναδικοί είναι ορισμένε ρυθμίσει, κανονιστικέ ρυθμίσει. Για παράδειγμα, ε, περιοχές που είναι ευαίσθητες στα αζωτούχα. Οι ανταγωνιστές μας έχουν τέτοια πράγματα. Το IPPC. Ε, αυτό είναι πονοκέφαλος για αυτούς που κάνουν εντατική εκτροφή ζώων. Και βέβαια δεν υπάρχει όφελος γιατί δεν μας επιτρέπουν να καλλιεργούμε γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς στην Ευρώπη, προϊόντα, ενώ παντού αλλού γίνεται. Και μετά επίσης δεν επιτρέπεται να θάβουμε τα ζώα θα χρειαστεί εγώ να πληρώσω άλλες 10.000 στερλίνες για να αγοράσω ε, ένα, ε, μια εγκατάσταση καύσεως για τα, για τα νεκρά ζώα. Και έχουμε και την οδηγία μετά ε, της, των ωραρίων εργασίας. Άλλος πονοκέφαλος αυτός. Και δεν υπάρχει αλλού. Ε, μετά η οδηγία για τα ζυζανιοκτώνα που για πολλές ε, μικρές καλλιέργειες δεν εξή τον κόπο να δημιουργούνται τα ζωνευτών αυτά, διότι έχουν κάνει τόσο δύσκολου του κανόνε τη καταχώρηση εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει νόημα. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τις ε, καλλιέργειε αυτέ και αναγκαζόμαστε να τις ε, εισάγουμε. Με άκουσαν άλλοι να μιλούν και για συστοιχίε κλοβών ορνήθων κλπ. Αυτέ έχουν απαγορευτεί εδώ αλλά όχι αλλού. Και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και χθιάλευρα, διότι έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την απίστευτη ε, ε, πολιτική της απόρριψης των ανεπιθύμητων ψαριών στη θάλασσα, νεκρών βέβαια, και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ηχθιάλευα. Ενώ αυτά δεν συμβαίνουν αλλού. Ρωτήσατε εσείς δύο πράγματα για το πρόβλημα του εισοδήματος των γεωργών. Η δύναμη των διαμεσαζόντων ή η αδυναμία των παραγωγών. Αυτό είναι μια τεράστια δυσκολία. Και μέσα στα χρόνια είδαμε τα μεγάλα σούπερ μάρκετ όπως Τέσκο κλπ. να έχουν αναπτυχθεί σε τεράστιο βαθμό. Ενώ οι αγρότες δεν έχουν γνωρίσει παρόμοια ανάπτυξη. Και έχουμε αυστηρούς κανόνες, έχουμε και την Επιτροπή Ανταγωνισμού κλπ που διασφαλίζουν ότι τελικά οι αγρότες δεν πρόκειται ποτέ να αναπτυχθούν διότι φοβούνται οι επιτροπές αυτές ότι θα βλάψουν τους καταναλωτές εν τέλει. Ίσως να μας πείτε εν τέλει τι νόημα έχει η στήριξη αυτή. Και εγώ πιστεύω είναι ότι είναι για να συνεχίσει να υπολειτουργεί η ε, γεωργία σε ε, ε, εποχές μεγάλων πλονασμάτων μία φορά, ένα χρόνο δηλαδή μπορεί να αποδώσει ένα εκτάριο, ένα τόνο ε, στάρι και του χρόνου να αποδώσει τέσσερις τόνους. Αυτά οφείλονται και στον καιρό. Και, και μετά ε, πέφτει μια ξηρασία στο νότιο ημισφαίριο και δεν υπάρχει ψωμί να φάει ο κόσμος. Πάντως σα ευχαριστώ εν τέλει για τη θαυμάσια παρουσίαση του θέματος. Ευχαριστώ κύριε Άγνιο. Στο Γιάννοφ. Πρόεδρε με μεγάλη χαρά άκουσα αυτά που είπε ο κύριος Άγνιου. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη γεωργία και επομένως μπαίνει και σε πολλές ε, λεπτομέρειες και σε συγκεκριμένα παραδείγματα που θα ήθελα και εγώ να θίξω. Η εντύπωσή μου από αυτά που ακούσαμε από την παρουσίαση είναι ότι ο προσκεκλημένος μας δεν επιθυμεί τις άμεσες πληρωμές. Είναι καταστροφικές, λέει, για την, για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ε, μίλησε για την, τις άθλιες αυτές άμεσες πληρωμές, για το κακό που κάνουν. Ε, Παρ' αυτά, υπάρχει ένα σημαντικό θέμα που συνδέεται με, με τις άμεσες πληρωμές και το ανέφερε και ο κ. Σάρνιο. Ποιο είναι οι διαφορετικές προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι Ευρωπαίοι γεωργοί σε σχέση με τις προϋποθέσεις και τους κανόνες που πρέπει να τηρούν οι υπόλοιποι γεωργοί του κόσμου. δεν συμφωνώ με το ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να τρώνε ασφαλή τρόφιμα και οι υπόλοιποι όχι. Υποτίθεται ότι δίνουμε βοήθεια στους Ευρωπαίους γεωργούς για να φτιάχνουν ε, πιο ποιοτικά τρόφιμα αλλά υπάρχουν και κάποια θέματα που δεν συνδέονται με την καλή ποιότητα των τροφίμων. Φερρυπίν η ευημερία των ζώων. Αν ζήσει και πεθάνει ευτυχισμένο ένα ζώο, ας πούμε, υποτίθεται ότι το προϊόν θα είναι καλύτερης ποιότητας, αλλά αυτό δεν είναι και σίγουρο στο κάτω-κάτω. Ποιο μα μας το λέει αυτό. Ε, δεν έκανε ποτέ καμία συνεδρίαση η η Επιτροπή μας για να συζητήσουμε τέτοια θέματα. Ε, και να σταθούμε και να τα αναλύσουμε. Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα του ΠΟΕ, και εδώ μπήκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα ο κύριος Σάγνιου. είναι πολύ γνωστό ότι κάθε χώρα επιδοτεί τη γεωργία της. Όλες οι χώρες το κάνουν. Επομένως, αν αρχίζουμε να κατηγορούμε ένα τον άλλον μέσα στον ΠΟΕ, αν αρχίσουμε να στυλιτεύουμε ο ένας τον άλλον για άνηση μεταχείριση, τότε δεν έχει τελειωμό αυτή η ιστορία, αυτές οι αλλοκατηγορίες. Αρχίζουν οι κατηγορίες της α χώρας εναντίον της β, της β εναντίον της γ, της β εναντίον της α και δεν λύνεται το πρόβλημα. Δεν μας βγάζει πουθενά αυτή η συζήτηση. Επομένως, Δεν νομίζουμε ότι το πρόβλημα έγκυται στον ΠΟΕ. Θέλω να πω όμως ότι τα συμφέροντα των Ευρωπαίων γεωργών δεν μπορούν να εξαρτώνται από αστάθμητους μελλοντικού παράγοντες. Δεν μπορούμε να λέμε ότι α, θα υπάρξουν συγκρούσεις στον ΠΟΕ και άρα εμείς θα κάνουμε αυτό. Όχι, εδώ είμαστε εδώ πέρα για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων γεωργών. Ε, πρώτα πρέπει να σκεφτούμε αυτά και μετά να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι μπορούν να πούν οι τρίτες χώρες οι, οι διεθνεί οργανισμοί. Γι' αυτό ακριβώ θέλω να κάνω ε, διάφορες ερωτήσεις στον ομιλητή μου. Είναι τόσο κακό αυτό το σύστημα των άμεσων πληρωμών. Έτσι μας είπε. Ούτως ή άλλως μόνο επικρίσεις ακούσαμε από αυτόν. Επομένως, αν δεν σας αρέσει αυτό το σύστημα, ποια είναι η εναλλακτική λύση στις άμεσες πληρωμές. Ποια άλλη πολιτική θα μπορούσε να αναπτύξει, να προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντικαταστήσει το σύστημα των άμεσων πληρωμών. Εν συνεχεία. Ρωτάω τον ομιλητή μας, ο οποίος επίσης ήταν πολύ επικριτικός για το πρασίνισμα, για τον, τη νέα συνιστόσα του πρασινίσματος του πρώτου πυλώνα και είπε μπορούμε να τη μεταφέρουμε στο δεύτερο πυλώνα. Αν ακυρώσουμε αυτή τη συνιστόσα, και να μην υπάρχει καθόλου. Τι γνώμη έχετε, θα ήταν καλό αυτό. Τρίτον, τι θα λέγατε για τα εισαγόμενα προϊόντα, τα οποία παράγονται με βάση λιγότερο αυστηρές προϋποθέσεις. Τι έχετε να πείτε για αυτά τα τρόφιμα. Ευχαριστώ, κυρία Στογιανόφ. Συνεχίζουμε τους ομιλητές μας. Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο κύριος Ολέινια Τσεκ. Εγώ δεν παίρνω το λόγο πολύ συχνά. Συνήθως είμαι ακροατής και όχι ομιλητής. Θα ήθελα να σας πω κύριε καθηγητά ότι στην Πολωνία όμως ήμουν υπουργό Γεωργίας επί δύο χρόνια ε, λίγο πριν ενταχθεί η Πολωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, γνωρίζω πολύ καλά τη γεωργική πολιτική και την ΚΑΠ, γιατί ασχολήθηκα με την σαφή μεταφορά της στην Πολωνία. Όταν ο καθηγητής μας έκανε την παρουσίασή του, τον άκουσα φυσικά, και μπορώ να συμφωνήσω με τα περισσότερα από αυτά που είπε. Όντως, θα πρέπει να δούμε αν η ΚΑΠ μας αρέσει ή όχι. Ιδίω ό,τι αφορά τι άμεσε πληρωμέ, αλλά όχι μόνο για αυτέ. Και για το δεύτερο πυλώνα. Μα αρέσει ο δεύτερο πυλώνα. όπου σε πολλές περιπτώσεις προσπαθούμε να υπερασπιστούμε κάποιες λύσεις με εργαλεία τα οποία σκοπό έχουν να χρηματοδοτήσουν συγκεκριμένες παραγωγές. Ένας από τους προλαλήσαντες μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται όταν ε, κατανέμονται διάφοροι πόροι στα διάφορα κράτη-μέλη. Δηλαδή παρατηρείται τότε μια τρομερή ανισότητα και αδικία για το ίδιο πρόγραμμα. Ακόμα και στο ίδιο κράτος μέλος υπάρχουν διστάμενες απόψεις. Ε, ακόμα και μεταξύ των γεωργών υπάρχουν διστάμενες απόψεις. Τώρα, η πρόταση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αλλάζει τίποτα ως προς αυτό. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δηλαδή, διατηρείται αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ των κρατών μελών και απεικονίζεται και σε όλα τα επίπεδα και τελικά φτάνει μέχρι τους ε, ε μεμονωμένους γεωργούς, όπου υπάρχουν διαφοροποίησεις μεταξύ αυτών. Αυτό είναι πρόβλημα. Από την άλλη, Προσπαθούμε να διατηρήσουμε την παραγωγή σε ορισμένες εκμεταλλεύσεις και σε περιοχές όπου οι άμεσες πληρωμές είναι σημαντικό τμήμα των εσόδων και των κερδών. Συνήθως αυτές είναι εκμεταλλεύσεις που δεν έχουν μεγάλο τζίρο, γιατί ακριβώς βασίζονται σε αυτό το σύστημα υποστήριξης, άμεσες πληρωμές δηλαδή. Και τελικά αυτό απεικονίζεται ε, σε απευθεία σχέση και στην τιμή του προϊόντος. Επομένως, υπάρχουν διάφορα επίπεδα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στην ΚΑΠ. Διάφορα στοιχεία. Έχουμε διάφορους ορισμούς, διάφορες παραμέτρους, αλλά το σύστημα παραμένει το ίδιο. Θέλουμε να σεβαστούμε τους κανόνες του ΠΟΕ, πρασίνισμα κτλ. Επομένως παίζουμε με τους ορισμούς, ε, τους αλλάζουμε αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Ακριβώς αυτό έλεγε και ο καθηγητής. Ε, το ίδιο ακριβώς είπε και ο Δανός Πρωθυπουργός. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε το greening ως στόχο ε, μια συγκεκριμένη εκμετάλλευση, αλλά θα πρέπει να είναι ο στόχο μια συγκεκριμένη περιοχή. Το ίδιο για τον ορισμό του ενεργού γεωργού, του, του ενεργού αγρότη. Δεν έχουμε αλλάξει τίποτα σε ό,τι αφορά το συνολικό πλαίσιο και σε λίγα χρόνια θα ξανααντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα με σήμερα με τη γεωργική παραγωγή. Γιατί δεν έχουμε αλλάξει επί τη ουσία τίποτα. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να βλέπουμε την ΚΑΠ όπω την αντιμετωπίζουμε σήμερα. Για μερικούς η ΚΑΠ είναι ένα είδος κοινωνικής επιδότησης. Δηλαδή ε, βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι λίγο κακομύριδες και που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Υπάρχουν γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα νέα κρατημέλη, όπου ο πληθυσμός είναι αρκετά φτωχός. Έχουμε μικρές λοιπόν γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Έχουμε ας πούμε μερικές οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις με πέντε παιδιά ας πούμε. Ε, από την άλλη έχουμε, μπορεί να έχουμε και τελείως διαφορετικές μη οικογενειακές ε, εκμεταλλεύσεις που όμως παίρνουν την ίδια στήριξη. Δεν είναι σωστό αυτό χρειαζόμαστε τεράστιες αλλαγές ε, ευρείας εμβέλειας. Καθηγητή, κύριε καθηγητά, σήμερα υπάρχουν και ακούγονται αυτές οι επικρίσεις. Υπάρχουν κάποιες επικρίσεις που δεν μπορώ να δεχτώ, ειδικά στο εσωτερικό αυτής της Επιτροπής. Ακούσαμε συχνά σε διάφορα κράτη-μέλη ότι η ΚΑΠ δεν είναι στο ύψος των προσδοκιών των γεωργών μας. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτές τις κριτικές που λένε ότι δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι αδικίες. Ξέρουμε ποιε είναι οι καταστάσει, ξέρουμε ποιε είναι οι αδικίες. Ας αλλάξουμε τα προβλήματα, τι προβληματικέ καταστάσει. Α αλλάξουμε τα προβλήματα. Στην πραγματικότητα προσπαθούμε να υπερασπιστούμε κάτι που τεχνικώς πώ δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε. Υπάρχει το θέμα του δεύτερου πυλώνα. Υποτίθεται ότι θέλουμε να βελτιώσουμε τη ζωή στις ε, περιοχές υπαίθρου. Παραδείγματο χάρη, έχουμε επενδύσεις για το ίντερνετ. Ε, δημιουργούμε, πράσινες, δημιουργούμε συγκεκριμένες μικρές εκμεταλλεύσεις με συγκεκριμένη λειτουργία Σύμφωνοι, σωστό αυτό. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τέτοιου μηχανισμού που θα μα ε, βοηθήσουν να βελτιώσουμε τη ζωή στην Ήπεθρο και την πρόσβαση των πληθυσμών αυτών στα δημόσια αγαθά. Και τα κρατημέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συζητήσουμε από κοινού όλα αυτά τα στοιχεία. Η έκθεση του καθηγητή είναι από τα καλύτερα έγγραφα που είδαμε τα τελευταία χρόνια στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω ακόμα μια φορά. Μάρτιν Όσλινγκ e και μετά συνεχίζουμε. Κύριε καθηγητά, μου οφείλω να ομολογήσω ότι δεν μπορώ να συμφωνήσω με τις ευχαριστίες. Με αφήσατε πραγματικά με ανοιχτό το στόμα. Το ίδιο ανοιχτό, με ανοιχτό το στόμα μένω όταν ακούω τον Άγνιου. Διότι δεν καταλαβαίνω τι, καλά, τι θέλετε να μας πείτε. Μας είπατε κατά επανάληψη ότι είστε οικονομολόγο και δεν έχετε ιδέα από γεωργία. Μήπως ήρθατε σε λάθος επιτροπή. Μήπως πραγματικά δεν έχετε ιδέα από γεωργία. Όταν λέτε ότι δεν έχουν σχέση με το εισόδημα όλες αυτές οι πληρωμέ, έχετε κοιτάξει καθόλου τις στατιστικές εισόδηματο των γεωργών. Στη Γερμανία, και που η Γερμανία δεν είναι και καμιά φτωχή χώρα, το μισό από το εισόδημα των Γερμανών γεωργών προέρχεται από μεταφορές εισοδήματο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν τα διαγράψω αυτά, τότε και οι Γερμανοί οι Γεωργοί θα έχουν κάποιο προβληματάκι. Και να μην πω τίποτε άλλο για άλλες χώρες. Μπορεί να είναι άσχημο αυτό, μπορεί να είναι δυστυχέ αυτό, αλλά είναι ένα γεγονό, το οποίο δεν μπορώ να αγνοήσω. Όταν λέτε επίση ότι οι λάθο άνθρωποι παίρνουν τελικά τα λεφτά, σωστό είναι αυτό. Αυτό προσπαθούμε εμεί να αντιμετωπίσουμε τώρα με την αναθεώρηση τη ΚΑΠ με περικοπές και άλλα να μην φτάνουν τα χρήματα στα λάθος χέρια. Βγάζετε από τη μέση και τον ενεργό Γεωργό εσείς ευθύς αμέσως. Καλά βέβαια πρέπει να το συζητήσουμε. Αναφέρατε και το πανεπιστήμιό σας το οποίο δεν θα έπαιρνε ε, εισοδηματική ενίσχυση για τις ε, αγελάδες που εκτρέφει. Δεν έχει όμως σχέση αυτό με τη συζήτηση που διεξάγεται αυτή τη στιγμή εδώ. Διερωτώ με, εν πάση περιπτώσει, ποιο σας κάλεσε να έρθετε εδώ για να μας πείτε πράγματα τέτοια, τα οποία βρίσκω ότι είναι άσχετα με τη συζήτησή μας. Μιλήσατε πολύ και για τον ΠΟΕ. Μήπως έχει προσφύγει καθημών κανένα στον ΠΟΕ κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ δεν έχω καμία τέτοια είδηση. Διότι αν πάει έτσι το πράγμα, τότε πολλοί πρέπει να πάνε στο εδόλιο του κατηγορουμένου ενώπιον του ΠΟΕ. Οι Ευρωπαίοι είμαστε από τους πιο συμμορφούμενους με την πολιτική μας σε σύγκριση με άλλες μεγάλες βιομηχανικές ε, χώρες. Δεν βλέπω λοιπόν για ποιο λόγο μιλείτε τόσο πολύ για τον ΠΟΕ. Γύρω στη Δόχα, ε, και τι έγινε. Δεν είναι καν επίκαιρο το θέμα. Έχουμε πολύ περισσότερα προβλήματα με, τα, με τις διμερείς συμφωνίες. Αυτά είναι τα προβλήματά μας και καλύτερα να μιλήσουμε για αυτά. Την προηγούμενη, το προηγούμενη χρονιά πήγαμε στις ΗΠΑ με την Επιτροπή μας να δούμε τι γίνεται εκεί και είπατε κι εσείς ότι θεωρείτε ότι η πολιτική μας, η αγροτική μας πολιτική θέλει να αποφύγει την αλλαγή των διαρθρώσεων, των δομών. Αυτό βρίσκω ότι είναι ιδεολογικά, ιδεολογική τοποθέτηση. Πήγαμε στις ΗΠΑ οι οποίες έχουν 700.000 εκμεταλλεύσεις και εξακολουθούν και λένε ότι 300.000 από αυτές τους περισσεύουν. Για φέρτε τα τώρα τα στοιχεία αυτά στην Ευρωπαϊκή Γεωργία που έχουμε 12,5 εκατομμύρια ενεργούς γεωργούς, τι πρόβλημα θα είχαμε τότε διαρθρωτικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τις, ευρωπαϊκέ με τις ευρωπαϊκές μας γεωργικές διαθώσεις, ναι, θέλουμε να τις υπερασπιστούμε. Αλλά κάνουμε και κάτι υπέρ της εικόνας αυτής της γεωργίας στην Ευρώπη, υπέρ της υπαίθρου και πολλές περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχαν πολύ διαφορετική εικόνα εάν δεν υπήρχε πια ενεργός γεωργία εκεί. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα όσα είπατε είναι καθαρά ιδεολογήματα ενός οικονομολόγου. Ας λέγατε από την αρχή ότι αυτά που κάνουμε εδώ σας φαίνονται ανοησίες. Αλλά να έρθετε να μας πείτε ότι στην ουσία εδώ δαπανούμε λεφτά τα οποία δεν θα έπρεπε να δαπανούμε, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εγώ θα προτιμούσα να κάνετε συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά από τέτοιες δεν άκουσα καμία. Προβήκατε σε δηλώσεις ενός επιστήμονα που με λίγα λόγια μας είπατε ότι εδώ η δουλειά που κάνουμε είναι περιττή. Αυτό δεν το δέχομαι. Ευχαριστούμε Μάρτιν. Ρίτα äh, Εγώ βέβαια τα πράγματα τα βλέπω τελείως διαφορετικά, ότι εκπλήσω κανέναν όταν τα λέω αυτά. Εγώ χαίρομαι για την ξεκάθαρη και ειλικρινή αντιμετώπιση του θέματος. Άλλωστε κάνατε και μια πρόταση. Είπατε ότι θα χαιρόσασταν να δείτε να μειώνεται ο πρώτος πυλώνας και να μεταφέρονται περισσότερα κονδύλια στον δεύτερο, ώστε εκεί να γίνουν πιο στοχευμένα προγράμματα που να διαμορφωθούν και πιο αποτελεσματικά. Εγώ το βρίσκω αυτό και πιο ε, έντιμο και πιο δημοκρατικό, διότι κινδυνεύουμε να προωθήσουμε μια αναθεώρηση, στην ουσία μοναδικό σκοπό, την διατήρηση των διαθρώσεων και που δεν έχουν μέχρι τώρα αυτές οι διαθρώσεις βοηθήσει τους γεωργούς. Προχωράμε λοιπόν σε μια λογαριθμική αύξηση των δαπανών και ε, από αναθεώρηση σε αναθεώρηση αυτές αυξάνονται. Το πρόβλημα για μένα είναι ακριβώς αυτό. Νομίζω ότι με την αναθεώρηση το μόνο που θα κάνουμε είναι να συνεχίσουμε τα ίδια. Να πετύχουμε δηλαδή τον στόχο να έχουμε γεωργούς που να λένε δεν μπορώ άλλο, δεν θέλω να συνεχίσω άλλο, διότι τελικά οι αγρότες είναι και επιχειρηματίες, δεν προσφέρουν υπηρεσίες καθαρά ως αυτός σκοπό στην κοινωνία. Έτσι, στην ουσία, με την πολιτική αυτή οδηγούμε σε αποξένωση των ε, αγροτών. Δεν μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε ένα ευχολόγιο που ωστόσο δεν είναι διατεθειμένη η κοινωνία να αποζημιώσει τους γεωργούς εφόσον το τήρουν. Και γι' αυτό θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντικό, όπως, είχε όπως είχα προτείνει και στην ε, πρώτη μου έκθεση, να τα κάνουμε αυτό μέσω του δεύτερου πυλώνα, με προγράμματα, με συμβάσεις, εφόσον οι αγρότες ε, με, τι με τις τους πληρούν κάποιες προσδοκίες της κοινωνίας, τότε να αποζημιώνονται γι' αυτό. Εδώ υπάρχουν και πολλοί αγρότες μέσα στην Επιτροπή μας. Εδώ αυτά παίζουν ρόλο και στι διαπραγματεύσει των τιμών. Να πρέπει να γνωρίζουμε, γνωρίζουν μάλωστε, μάλλον ποια, ποιες ακριβώς άμεσες ε, ενισχύσεις καταβάλλονται για την εκμετάλλευση και αυτά περνούν τελικά και στις τιμές η αναθεώρηση των τελευταίων χρόνων και οι ιδέε του Μαξάρη ήταν αρχικά καλές, αλλά δεν υλοποιήθηκαν και δεν οδήγησαν στον επιθυμητό στόχο. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ειλικρινεί και να πούμε ότι τώρα ειδικά σε περιόδους κρίσεω, πρέπει να έλθουμε σε, κάποια, σε μια έντιμη αγροτική πολιτική, ε, να πούμε ότι μέχρι τώρα δεν απέδωσε και α έχουμε το θάρρο να ξανασκεφτούμε τα πράγματα με ε, νέα νοοτροπία και όχι να καταπνίγουμε κάθε νέα σκέψη. Εάν απλώς αναπτύσσεται παραπέρα ένα μοντέλο το οποίο δεν λειτουργεί, τότε πραγματικά θα πέσει το κρεμό και δεν νομίζω ότι εξυπηρετούμε έτσι την Γεωργία. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ που καταστήσατε απόλυτα σαφές ότι υπάρχει και κάποια άλλη άποψη από αυτήν η οποία διατυπώνεται πάντοτε προς τα έξω. Και απλώς σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ, Μπρίτα. Μάριτ. before. Geht take it out. Wait, wait. Okay, you hear me now? Μ' ακούτε τώρα, ε? πριν δεν ακουγόμουν. Ωραία, άρα ξαναρχίζω από την αρχή. Να σας ευχαριστήσω. Καταρχάς διάβασα τις διαφάνειες ε, πριν ε, έρθω. Ε, δεν άκουσα όλη την παρουσίασή σας και ζητώ συγγνώμη, αλλά άλλο να είσαι ακαδημαϊκός και άλλο να είσαι πολιτικός. Νομίζω το καταλάβαμε και από την παρουσίαση. Ίσως ε, πριν από δύο χρόνια θα ήταν χρήσιμο να είχαμε ακούσει αυτή την παρουσίαση. Φοβούμαι όμως ότι τώρα είμαστε σε τελείως διαφορετική θέση. Δεν ξέρω αν ε, ε, άκουγα αυτή τη συζήτηση πίνοντας ένα ποτηράκι κρασί και τρώγοντας το δείπνο μου, ναι. Αλλά τώρα να, πρέπει να δούμε πώς θα τροποποιήσουμε την πρόταση που έχουμε μπροστά μας. Και μπορεί να ακούγομαι και κάπως εκνευσμένη, αλλά τι να κάνουμε. Να σας κάνω και την εξής παρατήρηση. Αν εγώ προσπαθούσα να βρω ένα ε, μηχανισμό στήριξης ε, και είμαι γεωργική οικονομολόγος, ε, δεν νομίζω θα το έκανα με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει μια σειρά μεταρρυθμίσεων της κοινής γεωργικής πολιτικής. Εμείς στην Επιτροπή μας προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά με μια δέσμη διαφορετικών μέτρων και περιορισμένο προϋπολογισμό. Έχω μελετήσει το νεοζηλανδικό, το αμερικανικό, το καναδικό μοντέλο που συζητήθηκε και εδώ και νομίζω ότι αυτό που έλειπα από την παρουσίασή σας ήταν το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά κάνει λόγο για εδαφική ισορροπία και αυτό είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους έχουμε αυτή τη στήριξη. Είναι πολύπλοκη γεωργία ε, αυτή τη θεωρία ε, treadmill theory την ξέρετε πράγματι. Οι αγρότες πρέπει να σας πω ότι δεν ελέγχουν ούτε τι παίρνουν ούτε ε, τι δίνουν για, τις, ε, για τα input. Και υπάρχει μια νέα διάσταση στην εξίσωση των δημόσιων, τα δημόσια αγαθά. Ήρθατε εδώ με μια αξία για τα δημόσια αγαθά που ίσω είναι πολύ ψηλότερο από τον προπλησμό που έχουμε για την κοινωνική πολιτική αυτή τη στιγμή και ίσω αυτό θα μα είχε βοηθήσει στη συζήτηση. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Αλλά οι μόνε σαφεί συστάσει που δίνεται είναι να περάσουμε ε, κάποια χρήματα στον ε, δεύτερο πυλώνα. Αυτό το είχαμε αποκλείσει, το είχαμε απορρίψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και η δεύτερη, σε ό,τι αφορά του ενεργού αγρότε, το είχαμε αποκλείσει και αυτό. Ε, και φαίνεται από την. Ε, συζήτηση. Εσείς ε, που θέλετε να την καταργήσετε αυτή την έννοια, πώς την, ε, με τι θα την αντικαταστήσετε. Οι Νεοζηλανδοί κατάργησαν μια ανοιχτή της επιδοτήσεις. Αυτό είχε πολύ δεινές επιπτώσεις και για τους αγρότες και για, τους, ε, και για τον τραπεζικό τομέα. Εμείς δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο και στη συζήτησή μας αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε. Εντάξει, να έχουμε και κάποια ακαδημαϊκή συζήτηση όπω αυτή τη στιγμή, θεωρητική συζήτηση, αλλά ο στόχος μας πιο πολύ είναι να τροποποιήσουμε μια πρόταση που έχει πολλού ε, σκοπού και την αναδιανομή, αλλά δεν θέλει να δημιουργήσει τριγμού στο σύστημα σε ό,τι αφορά την παραγωγή τροφίμων εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να επεκταθείτε λίγο περισσότερο πάνω στο πώ μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Έχω τις διαφάνειες σας εδώ, μιλάτε για τις επιπτώσεις ε, των άμεσων ε, πληρωμών λέτε ότι δεν θα επηρεάσουν ε, με διαρκή τρόπο τα εισοδήματα των αγροτών. Με τις κρίσεις που έχουμε βιώσει μέχρι τώρα υπήρχαν κάποια χρήματα τουλάχιστον για τη γεωργία. Κεφαλαιοποιούνται στις τιμές της γης. Και το τρίτο σημείο σας που λέτε ότι θα συνεχίσει να εξαρτάται πάρα πολύ από τις πληρώμες η γεωργία. Είναι τόσο σοκαριστικό αυτό, λέτε ότι είναι σοκαριστικό. Γιατί έτσι είναι και γιατί να έπρεπε να είναι αλλιώ. Τι θα πούμε στους ε, καταναλωτές ε, να πληρώσουν άμεσα περισσότερα πράγματα, όλα αυτά για τα οποία συζητάμε, δημόσια αγαθά. Εγώ είμαι κάπου στη μέση ε, μεταξύ χάουσλινγκ και άγνιου, αλλά αυτό που θα ήθελα αυτή τη στιγμή θα ήταν να μου δώσουν κάποια κατεύθυνση προς τα που να οδεύσουμε οι ακαδημαϊκοί. Αυτό θέλω να με βοηθήσουν πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ, Μαριάν. Ο Αντιπρόεδρος Σιακυριέσκη. Ευχαριστώ. Είμαστε σήμερα έχουμε 29 Φεβρουαρίου 2012. Ε, θα ξανά έχουμε 29 Φεβρουαρίου σε τέσσερα χρόνια. Δίσεκτο έτος. Ίσως γι' αυτό ακούγονται όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, ε, θέλω να ξεκινήσουμε μια ερώτηση προς τον καθηγητή. Στην ανάλυση σας, λάβατε υπόψη συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Γεωργίας ή βασιστήκατε μόνο ε, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Βρετανικής Γεωργίας λάβατε υπόψη σας τη διαφοροποίηση που υπάρχει στην ευρωπαϊκή γεωργία, στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής γεωργίας. Τι θα συνέβαινε χωρίς επιδοτήσεις, χωρίς υποστήριξη, χωρίς στήριξη της γεωργίας. Επίσης, άλλο ερώτημα. Η πολιτική. μπορούν να καταστήσουν όμοιρο μιας, ε, έναν τομέα της, ε, των εισαγωγών. Ε, Παραδείγματο χάρη ό,τι αφορά τον ε, ανεφοδιασμό μας σε τρόφιμα. Σκεφτείτε κάτι ένα παραλληλισμό με τον ενεργειακό ανεφοδιασμό. Υπάρχει περίπτωση κάποιος πολιτικός να αποφασίσει ότι εγώ θα καταστήσω την Ευρώπη όμοιρο, ας πούμε, των εισαγωγών. Θυμάστε την ε, κρίση των τροφίμων το 2007. Ευτυχώς η Ευρώπη δεν ε, πλήγηκε πολύ από αυτή την κρίση. Αλλά τότε, ακόμα και οι αρνητικοί ευρωβουλευτές, ακόμα και οι επικριτές της ΚΑΠ, αρχίσαν να λένε «Μα τι μπορούμε να κάνουμε στην ΚΑΠ, ούτως ώστε να μην ανησυχήσουμε ποτέ για τέτοιες ε, δυσκολίες, τέτοια προβλήματα ανεφοδιασμού σε τρόφιμα της Υπήρου μας». Της Υπήρου μας της μας σε ό,τι αφορά τις τιμές τώρα των γεωργικών προϊόντων, πού οφείλονται αυτές οι τιμές των γεωργικών προϊόντων, τα τις αναλύσατε στην παρουσίασή σας. Πώς καθορίζονται οι τιμές των γεωργικών προϊόντων. Ορισμένες από τις απόψεις σας ε, είναι δικαιολογημένες, αλλά μόνο μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αν λάβουμε υπόψη μας ορισμένα χαρακτηριστικά δηλαδή. Άκουσα και μια ενδιαφέρουσα θεωρία που εξέφρασε ο κύριος Ολένιτσεκ, πρώην υπουργό Γεωργίας. Αυτή τη θεωρία μπορείτε να την, να την ξαναπείτε στο πολωνικό κοινό, δημόσια. Είσαστε τόσο τολμηρός. Και πώς θα την ε, δεχόταν το κοινό, η Πολωνοί. Έτσι, Έχω αυτή την περιέργεια. Τέλος, καθηγητή. Στην Ευρώπη δεν έχουμε ένα πολύ διαφοροποιημένο σύστημα. Αν το θεωρήσουμε αυτό ως δεδομένο, με, αυτή... με δεδομένη αυτή τη διαφοροποίηση, τι απορρέει από αυτήν, τι μπορούμε να τροποποιήσουμε. Παραδείγματο χάρη για το greening, για το πρασίνισμα. Γιατί πρέπει να πληρώσουμε δύο γεωργούς τελείως διαφορετικά τον έναν από τον άλλον για το ίδιο πράγμα, για το πρασίνισμα. Για ποιο λόγο. Για την, το ίδιο πρασίνισμα, για την ίδια δραστηριότητα, γιατί πληρώνουμε τον α χ και τον β ψ. Όλα αυτά τα σημεία θα ήθελα να τα διευκρινίσουμε. Συγγνώμη. Ναι, ναι, ο κύριο Ολένιτσεκ. Έχετε δικαίωμα να απαντήσετε, βέβαια, Λίμωνο. Ε, τώρα θέλω να απαντήσω, όπω φαντάζεστε, στο φίλο μου εδώ πέρα, τον αντιπρόεδρο, με τον οποίο έχω συνεργαστεί χρόνια και χρόνια. Οι απόψει μου για την κοινή αγροτική πολιτική είναι γνωστές. Τις έχω εκφράσει κατ' επανάληψη. Έχω ένα φίλο ακαδημαϊκό που μου είπε ότι στους γεωργούς πρέπει να λέμε πάντα την αλήθεια. Γι' αυτό ακριβώς ε, με εκτιμούν οι γεωργοί γιατί πάντα μίλαγα έξω από τα δόντια. Πάντα έλεγα την αλήθεια για την ΚΑΠ και για τις επιπτώσεις της. Όλες αυτές τις θεωρίες που τις ακούσατε σήμερα μπορώ να τις πω ανα πάσα στιγμή και στο πολωνικό κοινό. Ίσως εσείς έχετε δυσκολίες και φοβάστε να μιλήσετε ανοιχτά στο κοινό. Μισελ Νταντάν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τα δικά ερωτηματικά, αγαπητέ κύριε καθηγητά, είναι διαφορετικά σε σχέση με αυτά που είπατε στην παρουσίασή σας. Επανειλημμένω, δείξατε ότι, ή τέλο πάντων δηλώσατε, ότι η κοινή γεωργική πολιτική δεν εξασφάλισε τελικά ένα εισόδημα μέχρι σήμερα αντίστοιχο με αυτό σε άλλους κλάδους. Και σίγουρα αυτό είναι αδιαφεσβητητό, αλλά ως οικονομολόγος ε, θέλω να μου πείτε, έχετε αποτελέσματα από κάποιες μελέτες ή προσωμιώσεις, εξομοιώσεις για το τι θα έχει γίνει η Γεωργία αν τα τελευταία 20 χρόνια δεν υπήρχε κοινή γεωργική πολιτική και η ενισχύση του πρώτου πυλώνα. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Αναφέρατε τη δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα. Και είπατε ότι τελικά ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που θέλει, να μπορεί να κάνει αυτό που θέλει. Πιστεύετε όμως ότι αυτό συνάδει τελικά με το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμεί να δημιουργήσει μια μεγάλη αγορά με όσο το δυνατόν πιο κοινούς κανόνες για όλους. Επόμενο ερώτημα. Πολλές φορές αναφερθήκατε στον ΠΟΕ. Σχεδόν ε, ε, αναφερθήκατε και στην περίπτωση αυτή του ΠΟΕ σαν μια απειλή. Ο κύκλος της Ντόχα για μένα πέθανε. Ο Μαξάρη πριν από 20 χρόνια σε έναν άλλο κόσμο, δηλαδή ίσως είχε ένα όραμα και ένα σχέδιο, αλλά αυτή την δεκαετία που πέρασε έχει αλλάξει ο κόσμος πιο πολύ από ό,τι όλον τον 20ο αιώνα. Είδαμε να αναδύονται νέες δυνάμεις, νέα ζήτηση, τίθεται εκ νέου και από διαφορετικού όρους ε, το γεωργικό ζήτημα και δεν έχει να κάνει μόνο με τη γεωργική παραγωγή, αλλά και με την παραγωγή τροφίμων. Αυτά μπαίνουν στο επίκεντρο, τα τρόφιμα, παραγωγή τροφίμων. Μήπως λοιπόν η δύναμη δεν έχει περιοδικά από τον ΠΟΕ μια εμπορικά, καθαρή, μάλλον εμπορική αμυγός τομή στο G20 και στη ΦΑΟ. Άρα δεν πρέπει να δούμε την κοινωνική πολιτική με ένα νέο διαφορετικό μάτι χωρίς πλέον να αναφερόμαστε στον ΠΟΕ που κλείνει τα 20 χρόνια που να είναι και που νομίζω ότι ετοιμάζεται να αφήσει τη θέση του στο διμερές και όχι στο πολυμερές σύστημα. Και να πω και κάτι άλλο. Το θέμα της διακύμωσης στον τίμο δεν το αναφέρατε. Είναι όμως ένα νέο φαινόμενο ή τέλος πάντων ένα φαινόμενο που γνωρίζει ε, πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις τελευταία. Πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους αγρότες με τα κονδύλια της ΚΑΠ να αντιμετωπίσουν αυτές τις διακοιμάσεις τιμές. Ευχαριστώ Μισελ. Καλυμνόφσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι άμεσες πληρωμές βρίσκουν σύμφωνους τους περισσότερους από εμά ως προς το ότι έχουν πολλά μειονεκτήματα. Συμφωνώ με τον καθηγητή που λέει ότι αυξάνεται και φουσκώνει η τιμή των γεών. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε επίσης για δίκαιη κατανομή των πόρων. Συμφωνώ με τον καθηγητή που λέει ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε το δεύτερο πυλώνα. Επίσης, στην Πολωνία έχουμε μια πολύ σημαντική, μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. Γιατί αν σκεφτείτε την κατανομή των πόρων ε, ανάμεσα στον πρώτο και στον δεύτερο πυλώνα, είμαστε στο 50-50. Υπάρχει ισοτιμία. Και από άλλες εμπειρίες που, έχω, που έχουμε, ε, μπορώ να σας πω ότι πολλά κονδύλια φτάνουν στους ε, κτηματίες και στους γεωκτήμονες και όχι σε αυτούς που ασκούν την πραγματική γεωργία. Και δεν, έχω, δεν συμφωνώ εδώ καθόλου με τον καθηγητή που λέει ότι η έννοια του ε, ενεργού γεωργού δεν έχει καμία σημασία. Γιατί τα λεφτά, τα κονδύλια της γεωργίας πρέπει να φτάνουν σε αυτούς που κάνουν το γεωργό, που είναι γεωργοί. Ακόμα και αν έχουν πάρα πολλά μειονεκτήματα οι άμεσες πληρωμές, αυτή η θεωρία των οικονομολόγων για τις άμεσες πληρωμές, σύμφωνα με την οποία οι άμεσες πληρωμές είναι το 50% του εισοδήματος των γεωργών, όλα αυτά εμείς τα απορρίπτουμε. Δεν τα συμμεριζόμαστε. Αν, ήταν, αν δεν υπήρχαν αυτές οι άμεσες πληρωμές, τι θα είχε συμβεί δηλαδή ή θα έπρεπε να είχαν αυξηθεί οι τιμές, δηλαδή τελικά τα τρόφιμα θα γινόταν απρόσιτα στην Ευρώπη, γιατί οι τιμές πρέπει να είναι τέτοιες που να επιτρέπεται να μπορούν να έχουν πρόσβαση οι καταναλωτές σε αυτά τα τρόφιμα ή αλλιώς θα υπήρχε τρομακτική συγκέντρωση της παραγωγής. Δηλαδή, παρά τα μειονεκτήματα των άμεσων πληρωμών, τελικά αυτές οι πληρωμές έχουν ένα σημαντικό ρόλο. Ήπιζα από αυτή την παρουσίαση να ακούσω κάτι παραπάνω για την δίκαιη κατανομή των πόρων. Ο καθηγητής μας είπε ότι αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε σε πολιτικό επίπεδο και να πάρουμε πολιτικές αποφάσεις. Εγώ έχω να σας κάνω μια γενική ερώτηση. Ένας Γεωργός, Βρετανός ας πούμε, ή Ισπανός, ή Πορτογάλος, που έχει μια παραγωγή που του αποφέρει 250 ευρώ ανά εκτάριο, πώς μπορεί να είναι ανταγωνιστικός απέναντι σε κάποιον που για την ίδια ε, επιφάνεια λαμβάνει 450-500 ευρώ. Γι' αυτό στο παρελθόν ε, στηρίξαμε τη θεωρία του Τσόλος ε, που έλεγε ότι οι άμεσες πληρωμές έχουν ένα ρόλο πολύ σημαντικό και πρέπει να διατηρηθούν. Ο κύριος Γιάρ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ βέβαια και για την διάλεξη. Την παρακολούθησα στο υπολογιστή μου στο γραφείο μου. Πάντως είναι σωστό να γίνει μια αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών. Βέβαια ο καθένας μπορεί να ασκήσει αγροτική πολιτική, μπορεί και να φιλελευθερωποιηθεί απολύτως η γεωρική πολιτική, αλλά νομίζω ξεχάσατε μια πτυχή. Η κοινή αγροτική πολιτική δημιουργήθηκε για να υπάρξει η αγροτική διάσταση και να παραμείνει ζωή στην Ήπεθρο. Αλλά δημιουργήθηκε επίσης και καθιδρύθηκε για να διασφαλίσει τη βασική διατροφή των πολιτών. Αυτό φαίνεται λίγο ε, άσχετο σήμερα, διότι όλοι έχουμε συνηθίσει τα σούπερ μάρκετ να είναι γεμάτα. Αλλά δεν ήταν πάντα έτσι. Άλλο παράδειγμα, πόσο μας ενοχλεί και πόσο μας κοστίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ανεξάρτητη ενεργειακά. Με το παράδειγμα αυτό μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο μεγάλη αξία έχει ότι τουλάχιστον είμαστε ανεξάρτητοι από εισαγωγές τροφίμων. Είμαστε αυτάρκης, ανεξάρτητοι, αυτόνομοι, αυτάρκης αν θέλετε και επομένως δεν, ε, δεν υποκύπτουμε και σε εκβιασμούς σε ό,τι αφορά την προμήθεια των βασικών ειδών διατροφής. Αν κάποια στιγμή αποφασίσουμε ότι δεν το θέλουμε και δεν το αποφασίσουμε εμεί εδώ, η κοινωνία θα πρέπει να το αποφασίσει, όποιο θέλει τότε να απελευθερώσει απολύτω την ε, Ευρωπαϊκή Γεωργία, τότε όμως παρετείται και από αυτή την πτυχή της ασφάλειας. Μπορεί να αναρωτηθεί κανείς τι θα κοστίσει όλη αυτή η υπόθεση τότε. Για την ώρα κοστίζει το όλον 27 δεκάρες του ευρώ ανά άτομο, ανά ημέρα. Αυτό είναι το κόστος της ασφάλειας τροφίμων. Εγώ θεωρώ ότι είναι εντάξει. Όποιος θεωρεί ότι δεν είναι εντάξει, να έρθει να μας το πει, να μας το εξηγήσει και να το δούμε. Αυτή λοιπόν η πρώτη μου ερώτηση. Το λάβατε υπόψη αυτό, την ασφάλεια δηλαδή προμήθειας τροφίμων. Μπορεί να ζήσει κανεί τρει εβδομάδε χωρί αυτοκίνητο, αλλά δεν μπορεί να ζήσει τρει εβδομάδε χωρί να φάει. Εμένα που είμαι και πολιτικός που ασχολούμαι με την αγροτική πολιτική και που ίσως λέω ότι δεν τα έχουμε εξηγήσει αρκετά, η κοινή αγροτική πολιτική και ο Ευρωπαίος αγρότης εμφανίζονται συχνά ως αντίθετη με κάθε αλλαγή. Από το 1990 είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω ενεργά στην κοινή αγροτική πολιτική και μπορώ να πω ότι οι αγρότες οι μεταρρυθμίσεις, οι αναθεωρήσεις και όλες οι αλλαγές που έχουν υποστεί και έχουν ανεχθεί, κάθε τρία χρόνια έχουμε αναθεωρήσει την αγροτική πολιτική. Με πιο επιχειρηματική διάσταση, με πιο περιβαλλοντική διάσταση κλπ. Έχουμε ωστόσο μια πρώτη επιτυχία, δεν έχουμε πλέον σχεδόν επιδοτήσεις εξαγωγών, μεγάλη επιτυχία. Στην αρχή της αγροτικής πολιτικής οι μισές δαπάνες ήταν επιδοτήσεις εξαγωγών. Δεν έχουμε πλέον τέτοιες τώρα και έχουν γίνει και πιο φθηνά τα, ε, και είναι και πιο φθηνή η αγροτική πολιτική. Είπα 27 δεκάρες σήμερα, μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν 35 λεπτά του ευρώ ανά άτομο, ανά ημέρα, το κόστος της ΚΑΠ. Εμείς είμαστε εδώ στην πολιτική αυτή για να συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις. Έχουμε μια αφετηρία και έχουμε και ένα στόχο και σας παρακαλώ να μας δώσετε ίσως κάποιες υποδείξεις για το πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε καλύτερα και δικαιότερα και αποτελεσματικότερα την κοινή αγροτική πολιτική. Τελευταία παρέμβαση, ο Άλμπερτ. Ευχαριστώ, Άλμπερτ επίτηδες ζήτησα τελευταίο το λόγο γιατί ήθελα να ακούσω τις παρεμβάσεις των άλλων συναδέλφων. Κύριε καθηγητά, ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι δηλώσεις σας, ορισμένες μπορεί να με βρουν σύμφωνο, σε άλλες όμως είμαι υποχρεωμένο να προβάλλω ένσταση. Για παράδειγμα, ΠΟΕ, δεν ξέρω πού έχουμε φτάσει, σε, έχω, έχω πάει σε ορισμένες αγροτικές περιοχές του κόσμου, όπως και άλλοι συναδελφοί μου. Και όταν βλέπω την ληστρική καλλιέργεια που γίνεται σε ορισμένες περιφέρειες, τότε χαίρομαι που στην Ευρώπη έχουμε μια πολύ διαφορετική αγροτική πολιτική. Πήγα και στις Ηνωμένε Πολιτείες και φεύγοντας από τη Νέα Υόρκη να πετάξω στο Λος Άντζελες, είδα στην Καλιφόρνια κύκλους οι οποίοι την διάρκεια της ε, σποράς ήταν καφέ γιατί ρώτησα τους αγρότες είναι καφέ το χρώμα αυτών των μεγάλων κύκλων, διότι μου είπαν αρδεύουμε όλο και βαθύτερα, 50 μέτρα βαθύτερα από ό,τι πριν από 20 χρόνια και δεν, δεν προσέξαμε ότι αρχίσαμε να αντιλούμε αλμυρό νερό και επομένως τις αρδεύσαμε με αλμυρό νερό τις περιοχές αυτές και καταστράφηκαν. Τέτοια πράγματα λοιπόν δεν θέλω να συμβούν και εδώ. Μπορώ να σας πω και άλλα παραδείγματα από την Ινδία και την Κίνα που ε, σημειώνονται παρόμοιες εξελίξεις. 40% των διεμητριακών αυτή τη στιγμή αρδεύονται από βαθιά υπόγεια ύδατα. Προδεκαετίας είχα πάει στη Βραζιλία και έχω ξαναπάει πολλές φορές. Είχαμε πάει στην κεντρική Βραζιλία στην Λίνα που είναι μεγάλα ε, αγροτικά μεγάλες ε, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και εκεί αντλούνται τα νερά του ποταμού Ρεσίφε και η παραποτάμια πόλη Ρεσίφε δεν έχει πλέον νερό. Τι θα μας λέγατε εάν οι Ευρωπαίοι αγρότες τραβούσαν τα νερά του Δούναβη και τον αδειάζανε. Δεν είναι αυτή η αγροτική πολιτική που θέλουμε εδώ. Και επειδή η ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική έχει πολύ περισσότερα καθήκοντα, περισσότερες αποστολές και περιβαλλοντικές και επειδή η γεωργία γίνεται κατά βάση με τρόπο βιώσιμο. Για τον λόγο αυτό θεωρώ ένα ποσό ότι πρέπει να δίνεται ως αντιστάθμιση από τον πρώτο πυλώνα. Για το ύψος αυτής της αντιστάθμισης μπορούμε να συζητήσουμε. Έχω και ένα δεύτερο σχόλιο. Ποιε είναι δηλαδή οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι Ευρωπαίοι Γεωργοί. Έχω πει το παράδειγμα αυτό και άλλες φορές, αλλά εσείς βέβαια δεν ήσασταν παρόν αγαπητέ κύριε καθηγητά. Στις 27 Εβδόμου, 1961. Πήρα το δίπλωμα οδηγήσεως. Μία γερμανική τότε εφημερίδα είχε γράψει ότι κόστιζε τότε 5 λεπτά η εφημερίδα και ένα κιλό ε, δημητριακά κόστιζε 25 ε, σεντ. Σήμερα η εφημερίδα αυτή κοστίζει το 4,80 πλάσιο, ωστόσο τα, το κιλό των Δημητριακών κοστίζει λιγότερο από ό,τι κόστιζε τότε. Εάν είχε πάρει την ίδια ε, αύξηση θα έπρεπε σήμερα να κοστίζει 300, 350 λεπτά, δηλαδή 3,5 ευρώ το κιλό τα Δημητριακά. Τα ίδια ισχύουν και αλλού. Εάν λοιπόν υπολογίσω και 300 ευρώ φτάνω στα 1072 ευρώ και επομένως εξακολουθώ να βρίσκομαι πάντα κάτω από τον μέσο όρο απόδοσης του στρέμματος προ 50 ετών. Τι θέλω να πω. Αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας, καθώς επίσης με μεγάλο κόπο και μόχθο των αγροτησών και των αγροτών απέδωσε η Ευρωπαϊκή Γεωργία έτσι ώστε οι καταναλώτες και οι καταναλωτές να έχουν σήμερα φθηνά τρόφιμα στο τραπέζι τους χωρίς ταυτόχρονα να έχουμε καταλυστέψει την φύση. Αυτό που θα με ενδιέφερε και έχουμε στο τέλος της παρεμβάσεώς μου είναι να μας πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα πώς θα φανταζόσασταν την κοινή αγροτική πολιτική. Αυτό θα μας ενδιέφερε αν θέλετε να μας πείτε δηλαδή λίγο πιο συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τον καθηγητή. Ε, θέλω να μας κρατήσετε ξύπνιους. Τα καταφέρατε κύριε καθηγητά, διότι η συζήτηση ήταν τόσο ζωντανή και τόσο ενδιαφέρουσα. Τώρα, μπορώ να σας ξαναδώσω το λόγο κύριε καθηγητή, αλλά σας ζητώ να μας κάνετε και συγκεκριμένες προτάσεις. Γιατί έχουμε μπροστά μας επιτάπητος την νέα πρόταση για την ΚΑΠ. Και είμαστε εδώ πέρα για να πάρουμε αποφάσεις. Πρέπει να ψηφίσουμε αλλαγές, τις αλλαγές. Οι συγητέ μας είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν και μάλιστα μέσα σε σφιχτές προθεσμίες. Σας δίνω το λόγο, σας ευχαριστώ και σας ζητώ να χρησιμοποιήσετε αυτό το χρόνο για να βοηθήσετε την Επιτροπή μας ε, να πάρει αποφάσεις. Ευχαριστώ. Να προσπαθήσω. Πολύ ευρία, πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Να πω ευθύ εξ αρχής ότι είμαι οικονομολόγος, δεν είμαι πολιτικός, πάντα οικονομολόγος ήμουνα και έχω μεγαλύτερη ευχέρεια να οικοτολογήσω πάνω σε διάφορες υποθέσεις. Ε, Υπάρχουν μια σειρά από εργαστήρια που οργανώνεται επί των προτάσεων της Κομισιόν και εμένα μου ζητήσαν να μιλήσω για τις άμεσες πληρωμές. Ε, ακούστηκαν στη συζήτηση αυτή διάφορα άλλα θέματα, αλλά θα συζητηθούν σε άλλα εργαστήρια, όχι στο δικό μας. Εγώ μιλάω για τις άμεσες πληρωμές. Μου ζήτησαν λοιπόν να παρουσιάσω αυτή την έκθεση και μου είπαν ότι ο προσανατολισμός ε, θα πρέπει μάλλον να προσανατολιστώ ε, λαμβάνοντας υπόψη και τον ΠΟΕ, γιατί είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Παρότι συμφωνώ με πολλά σχόλια ότι ο γύρος της Ντόχα ε, πεθαίνει, εκπνέει και κάποια θέματα για την συμβατότητα των, α, των άμεσων πληρωμών με, με τον ΠΟΕ είναι ίσως καθαρά ακαδημαϊκά. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ασήμαντος ο ΠΟΕ. Αλλά είμαστε εκτό, εντός του συστήματος του ΠΟΕ, δεν είμαστε εκτός και με βάση τι συμφωνίε του ΠΟΕ που εξακολουθούν να είναι ενισχύ, ακόμη αν ας πούμε, επειδή είμαστε αυτό το σύστημα, αν τα άλλα έθνη ε, εκνευριστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική της, μπορεί να βρουν τρόπους για να προσφύγουν αντίον μας. Ε, Φερρυπίν με την πολιτική ζάχαρης. Ελπίζω να μην ήμουν πολύ προκλητικός. Παρ' όλα αυτά, ορισμένοι από εσά θεώρησαν ότι είμαι. Και ότι ε, ήταν σαφέ ότι είμαι οικονομολόγος. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι το σύστημα άμεσων πληρωμών αφορά α, μια ευρία γκάμα προϊόντων και συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε ένα ενίο σύστημα το οποίο να αντιμετωπίζει κάθε περιοχή, κάθε γεωργό ε, δίκαια, όταν είναι ενιαίο το σύστημα. Αυτή η λέξη δικαιοσύνη ακούστηκε πολλές φορές. Ως προς το ποσά που παίρνει ο κάθε γεωργός, και συμφωνώ με αυτούς που είπαν ότι δεν είναι δίκαιο το σύστημα και φυσικά σας είπα από την αρχή ότι ως οικονομολόγος δεν ξέρω πώς πρέπει να αντιμετωπίσω αυτή την δικαιοσύνη. Ε, ας πούμε, ο αριθμός των ευρώ είναι εκτάριο, Φερρυπίν. Θα μπορούσε να ένα μέτρο, ένας μπούσουλος. Αυτό όμως σημαίνει ότι οι μεγάλοι κτηματίες ε, εισπράττουν πολύ περισσότερο από τους μικρούς ε, εκμεταλλευτές. Του μικρού γεωργού. Επομένω, μπορεί να γίνει πολύ έντονη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Επίση, η λέξη δικαιοσύνη χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια του ανταγωνισμού. Δίκαιο ανταγωνισμό. Επανερχόμαστε σε αυτή την ιδέα του τι είναι οι άμεσε πληρωμέ. Αν είναι αποσυνδεδεμένε, τότε δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τον ανταγωνισμό. Αν οι άμεσε πληρωμέ είναι αποσυνδεδεμένε, δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τον όγκο της παραγωγή. Επομένω, το θέμα τη ε, ασφάλεια των τροφίμων δεν θα πρέπει να εκφεύγει ε, τη συζήτηση για τις άμεσες πληρωμέ. Αν πιστεύουμε ότι είναι σημαντικές για την ε, επιστηστική ασφάλεια, και αυτό είναι μια σημαντική προσδοκία, θα πρέπει να ξανασκεφτούμε όλο το σύστημα των άμεσων πληρωμών και πώς ε, ε, επηρεάζονται οι εμπορικοί μας εταίροι λόγω αυτού. Νομίζω ότι έκανα και κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Πρότεινα... Μη είπα μάλλον ότι δεν μ' άρεσε αυτή η πρόταση για τους ενεργούς ε, γεωργούς για δύο λόγους. Ε, ορισμένοι μπορεί να πιστέψουν ότι υπάρχει και ένα τρίτο λόγω τη σχέση με το Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ. Αλλά δύο λόγοι είναι οι βασικοί. Γιατί περιπλέκει τη σχέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ΠΟΕ, πρώτον. Και δεύτερον, γιατί καλύπτει πολύ διαφορετικά γεωργικά συστήματα που όλα αυτά μπορεί να επηρεάσουν δυνητικά την πολυλειτουργικότητα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Και μου φαίνεται ότι είναι σημαντικό ότι αν λέμε ότι η πολλαπλή συμμόρφωση και οι καλές ε, περιβαλλοντικές ε, της γεωργίας και το πρασίνισμα είναι σημαντικές προϋποθέσεις, τότε είναι παράλογο κατ' εμέ να αποκλείσουμε κάποιους διαχειριστές γης ή κτηματίες γιατί δεν είναι ενεργοί γεωργοί. Σα είπα επίσης ότι μια και η Κομισιόν πρότεινε ότι το 30% του προπολογισμού θα πρέπει να πάει σε αυτό το στοιχείο του πρασινίσματος, ίσως θα πρέπει να πάτε ένα βήμα παραπέρα. Για δύο λόγους πάλι. Ο πρώτος, γιατί πιστεύω ότι προς το παρόν η σύνδεση των αμέσων πληρωμών, ε, μάλλον των, βασικών πληρωμών με το πρασίνισμα, μέσω από το σύστημα, μέσω από το σύστημα του πρασινίσματος, όντως δημιουργεί προβλήματα στον ΠΟΕ και δεύτερον γιατί Πραγματικά πιστεύω ότι ένα σύστημα καταποκοπή, ένα ενιαίο μονοκόμματο σύστημα, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξοδέψουμε πολλά λεφτά, για να βελτιώσουμε το κριτήριο του πρασινίσματος, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Καλύτερο θα ήταν να βάλουμε αυτά τα λεφτά στο δεύτερο πυλώνα ή να πούμε, ναι, στον πρώτο πυλώνα ε, να παραμείνει εκεί, αλλά το διαχωρίζουμε το βασικό εισόδημα, τη βασική πληρωμή από το πρασίνισμα. Τα διαχωρίζουμε αυτά τα δύο. Και δίνουμε μεγαλύτερη ελευθερία στα κράτη-μέλη για να καθορίσουν αντικειμενικά κριτήρια για συγκεκριμένες περιοχές που θα πρέπει να πληρεί η συνιστός αυτού του πρασινίσματος. Κάτι που δεν είπα στην παρουσίαση αλλά υπάρχει στην έκθεση είναι ότι ένα χρήσιμο στοιχείο των άμεσων πληρωμών μπορεί να είναι η εδαφική συνοχή για την οποία γίνεται λόγος. Και θα μπορούσε οι άμεσες πληρωμές να δίδονται μέσα σε ένα πρόγραμμα περιφερειακής βοήθειας ε, που υπάρχει στο πράσινο κουτί. Με δεδομένη την πρόταση της Κομισιόν μπορούμε να βρούμε κάποια θετικά ε, μπορούμε να βελτιώσουμε κάποια άλλα, δεν είναι όλα αρνητικά. Δεν ήρθα εδώ με μοντέλα του τι θα συμβεί αν δεν υπάρξει καμία στήριξη της ευρωπαϊκής ε, γεωργίας. Δεν μ' να δουλεύω με μοντέλα, αλλά συμφωνώ με αυτούς που είπατε ότι αν αυτό κάναμε μία νυχτή θα ήταν καταστροφικό. Σας προτείνω λοιπόν να γίνουν κάποιες μικρές αλλαγές στην πρόταση της Κομισιόν. Αν με ρωτήσετε με τι θα πρέπει να μοιάζει η μελλοντική ΚΑΠ, θα απαντούσα ότι δεν είμαι σίγουρος ότι είναι σωστό το να συνεχίσουμε το σύστημα των άμεσων πληρωμών, γιατί αυτό σημαίνει ότι δρέπουν τα περισσότερα ωφέλη οι μεγάλοι κτηματίες, ε, το κόστος του όλου συστήματος. Αν θέλουμε να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο, τότε θα πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα βαθμιαίο που θα εφαρμοστεί ε, μέσα σε πολλά χρόνια. Και πριν από 20 χρόνια ε, ο καθηγητής Τάγκεμαν πρότεινε μία πλήρη αποσύνδεση του συστήματος μέσα σε μία 15ετή περίοδο, το λεγόμενο bond scheme. Ίσως θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε αυτό το σύστημα. Για το υψηλότερο κόστος που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι γεωργοί σε σχέση με τους υπόλοιπους γεωργούς του πλανήτη, όντως είναι πρόβλημα, το ομολογώ, για την επιστημιστική ασφάλεια. Όντως, θα πρέπει να ρυθμιστεί μέσα από κανονισμού για την επιστημική ασφάλεια. Επίση, είναι πολύ προβληματικό για την ευημερία των ζώων, αλλά σε ό,τι αφορά τα άλλα περιβαλλοντικά θέματα, θα έλεγα, ε, για μια στιγμή είμαστε ένα τμήμα του πλανήτη που με πυκνή έτσι πυκνοκατοικημένο και ούτως ή άλλως έχουμε και πολύ σημαντικούς δασμούς σε πολλά α, γεωργικά προϊόντα. Ε, η, τα σιτηρά και η ελαιούχοι σπόροι είναι εξαίρεση. Και η λογική ότι οι άμεσες πληρωμές υπάρχουν για να αντισταθμίσουν και να αποζημιώσουν τους γεωργούς για το υψηλότερο κόστος, αυτό σημαίνει ότι το σύστημα πληρωμής είναι διπλό. Γιατί αν παίζουν αυτό το ρόλο οι άμεσες πληρωμές, τότε χρειαζόμαστε τόσο ψηλούς δασμούς ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή το ένα κρατήστε ή το άλλο. Ή τι άμεσε πληρωμέ ή του δασμού. Αλλά έχουμε και τα δύο. Τέλο πάντων, τώρα αρχίζω να ξεπερνάω το πλαίσιο μέσα στο οποίο έπρεπε να κινηθώ ε, σήμερα, που ήταν να σχολιάσω τι προτάσει τη Κομισιόν για τι άμεσε πληρωμέ. Είμαι σίγουρο ότι ξέχασα κάποιε ερωτήσει, αλλά ε, αυτά είδα εδώ πέρα μπροστά να έχω σημειώσει, αυτά απάντησα. Ευχαριστώ τον καθηγητή. Και πάμε γρήγορα στο σημείο 14 της ημερήσιας διάταξης, τροποποίηση του κανονισμού 73 του 2009 του Συμβουλίου για την εφαρμογή των άμεσων πληρωμών στους γεωργούς ε, το 2013. Πρέπει να εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης που είχε παρουσιάσει ο Λούις Κάπουλα Σάντος για την εφαρμογή των άμεσων πληρωμών στους γεωργού για το 2013. Για... Όπως ξέρετε, ο σημερινό κανονισμός για τις άμεσε πληρωμές θα εξακολουθήσει να ισχύει και το 2013. Αλλά υπάρχουν κάποιες διατάξεις ε, χρηματοδοτικές ε, μέσα στον κανονισμό που λειτουργούν και θα ισχύσουν μόνο μέχρι το 2012. Επίσης, τα αιτήματα ενισχύσεων για το 2013 αφορούν το οικονομικό έτος 2014 τότε ο προπολογισμό της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ε, ενταχθεί σε ένα διαφορετικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, αυτή η πρόταση έγινε από την Κομισιόν για να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές διατάξεις για τη μεταβατική αυτή περίοδο, δηλαδή πριν από την υιοθέτηση της νέας ΚΑΠ. Ο Λούις δεν είναι εδώ μαζί μας, γιατί έχει ένα προσωπικό πρόβλημα, δεν είναι διαθέσιμος. Η Ράτσα όμως, Γκαρσία Πέρες, τον αντικαθιστά. Η Ράτσα έχει το λόγο. Υπενθυμίζω σε όλους τους συναδέλφους ότι μπορείτε να καταθέσετε τροπολογίες μέχρι τις 29 Μαρτίου, 12 το μεσημέρι. Ο, ο εισηγητής δεν έχει παρουσιάσει καμία τροπολογία, θα μας τα επιβεβαίωσε όλα αυτά η Ράτσα. El reglamento Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κανονισμός 73-2009 της ε, άμεσες πληρωμές που είναι σε ισχύ αυτή τη στιγμή έχει σε ένα παράρτημα πίνακες κατανομής ε, για τις άμεσες πληρωμές μέχρι το 2012. Για τα κρατημέλη θα πρέπει λοιπόν να δούμε τα ποσά ε, τα, στο πλαίσιο του δημοσιονομικού πλαισίου αλλά και για το προσεχές δημοσιονομικό έτος για το 2013 για τα γεωργικά έτη, επειδή είναι ιδιαίτερο και για τον γεωργικό προπολογισμό. Το 2013 είναι ε, ουσιαστικά τότε χρηματοδότηση το 2014. Η πρόταση της Κομισιόν για το 2013 προϋποθέτει παράταση ε, των ε, εθνικών ποσών του 2012 με κάποιες προσαρμογές που στόχο έχουν αφενός ε, να είναι σαφής ο μεταβατικός χαρακτήρας του έτους 2013 σε διαφορετικά δημοσιονομικά ρυθμιστικά πλαίσια για την κοινή γεωρική πολιτική και να εγγυηθεί επίσης την συνέχεια των τρεχόντων επιπέδων των άμεσων πληρωμών λαμβάνοντας υπόψη τις επιπλέον ανάγκες ε, για το phasing in ε, των προ, ε, πρόσφατων κρατών μελών και σε ό,τι αφορά επίσης και την εθελοντική διαφοροποίηση. Θέλω να ευχαριστήσω οι εισηγητή τη υπηρεσία Κομισιόν για τη διαθεσιμότητά του σε όλα τα στάδια της διαδικασία και καλό θα ήταν να γίνει μια συνάντηση για να διευκρινιστούν τα ασαφή σημεία και να απαντηθούν τα ερωτήματα. Θέλω επίση να τονίσω εξ ονόματο του εισηγητή τη σημασία που έχει να εγκριθεί γρήγορα αυτό ο κανονισμό και παραμένω στη διάθεσή σα για να ακούσω τι έχετε να πείτε ε, σε σχέση με έναν συνολικό συμβασμό στον οποίο θα μπορούσαμε να καταλήξουμε για να σεβαστούμε τις προθεσμίες αλλά να μην θέσουμε και σε κίνδυνο την καταβολή των πληρωμών στους αγρότες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλει κανένα να πάρει το λόγο για το σημείο αυτό. Αν όχι, κρατάμε τις παρατηρήσεις του εισηγητή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο. Sí. Prego. Παρακαλώ. Κομισιόν. Και ίσως μετά ακούσω και συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω πολύ απλά να πω ότι όπως ε, προείπε και η εισηγήτρια... Η πρόταση της Κομισιόν βέβαια είναι να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος άμεσων πληρώμων που προτείνει στο ίδιο πακέτο η Κομισιόν εφαρμόζεται από το 2014 και μετά δηλαδή οικονομικό έτος 2015. Επομένω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό που πολύ απλά προσπαθεί να κάνει είναι να εξασφαλίσει ε, ότι δεν θα αλλάξει κατάσταση για τις εφαρμογές το 2013 να ισχύσουν τα ίδια με το 2012 δηλαδή αλλά όπως νομίζω ότι έχει υποθεί και προηγουμένως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το phasing out και τα σχετικά ποσά για τα 12 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη και τα σχήματα τα οποία λήγουν το 2013, οικονομικό έτος 2013. Προερωτική διαφοροποίηση, μεταφορά κάποιων μη δαπανηθέντων πόρων στην έπτυξη τη υπαίθρου. Αυτά λοιπόν ε, θέλουμε να μεταφερθεί ό,τι ισχύει το 2012 και για το 2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να έχουν εγκριθεί τα μέτρα μέχρι το καλοκαίρι, γιατί από 1η Πρώτου 2013 θα έχουμε τον κανονισμό και θα πρέπει να ξέρουν οι αγρότες συγκεκριμένα τι ισχύει όταν θα καταθέσουν τα αιτήματά τους για το 2013. Ωραία δεν θέλουμε να πάρουμε το λόγο εμείς από πλευράς ευρωβουλευτών. Μπορούμε να συνεχίσουμε τάχιστα. Αν δεν υπάρχουν τροπολογίες, έχουμε μέχρι τις 22 Μαρτίου, μου λέει η Γραμματεία. Τελευταίο σημείο στη μέση διάταξη. Σημείο 15. Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά. Ο εισηγητής, ο αντιπρόεδρος κ. Βασεβόσκη θα κάνω μια ανταλλαγή απόψεων για την ε, ευημερία των ζώων, ιδίως κατά τη μεταφορά. Η Κομισιόν τον Νοέμβριο ετοίμασε μία έκθεση για την επίπτωση της ισχύουσας νομοθεσίας στην στο εσωτερικό εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ευημερία των ζώων κατά τη μεταφορά και στις ε, κοινωνικές επιπτώσεις της νομοθεσίας ε, εμείς ε, έχουμε μία έκθεση πρωτοβουλίας. Ο Αντιπρόεδρος θα κάνει την παρουσίασή του. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. No, pracujemy nad sprawozdaniem. E, e, prace przebiegają do... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχουν γίνει ήδη κατ' επανάληψη συναντήσεις για το θέμα. Ε, υπάρχει ένα πρώτο σχέδιο της ε, εκθέσεως. Οι βασικές, οι θεμελιώδεις διαπιστώσεις εν ώψη και των προτάσεων που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι ναι μεν υπάρχει κάποια πρόοδος σχετικά με, τους, με τις συνθήκες μεταφοράς, ωστόσο η πρόοδος αυτή δεν είναι επαρκής. Κυρίως όμως δεν έχει επιτευχθεί ένας εκ των κυρίων στόχων του κανονισμού του 2005 για, τους, για τις συνθήκες μεταφοράς ο στόχος δηλαδή της μείωσης του συνολικού αριθμού μεταφερόμενων ζών των ζώων. Από την έκθεση της Κομισιόν και μέχρι το 2009 διαπιστώνεται ότι υπήρξε σημαντική αύξηση των μεταφορών. 8% των χοιρινών, 6% των ε, προβάτων και μόνο για τα άλογα μειώθηκαν περίπου 17% τα μεταφερόμενα ζώα. Άρα, ο στόχος που είχε τεθεί το 2005 να, να μειωθούν δηλαδή οι μακρινές μεταφορές ζώων προς, ζών των ζώων που προορίζονται προσφαγή, φαγή. Δυστυχώς αυτός ο στόχος δεν επιτεύχθηκε. Η έκθεση τονίζει ότι οι μεταφορές, οι μακρινές μεταφορές προκαλούν κόστος αλλά και οικονομικό και κοινωνικό και ε, περιβαλλοντικό διότι αφενός βρίσκονται περισσότερα οχήματα στους δρόμους άρα περισσότερες εκπομπές καυσαερίων αλλά σημαίνει επίσης και ότι επηρεάζεται δυσμενώς η τιμή του κρέατος και των προϊόντων κρέατος το οποίο δεν αξιολόγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε μοναχά ότι οι μακρινές μεταφορές αυξάνουν το κόστος για τις επιχειρήσεις. Αλλά δεν ε, υπάρχει συνολική αποτίμηση όλου του κόστου, του συνολικού κόστους, διότι κάποιος επομίζεται το κόστος αυτό. Και εδώ μιλούμε καμιά φορά για χιλιάδες χιλιόμετρων. Τελικά το ε, βάρος του κόστους αυτού επομίζεται ο τελικός καταναλωτής είναι προφανές. Προτιμητέα θα ήταν η μεταφορά του κρέατος ή των προϊόντων κρέατος και όχι των ζώων των ζώων. Και κυρίως πρέπει βέβαια να τονωθεί η επιτόπου κατανάλωση, δηλαδή η παραγωγή, η σφαγή κατανάλωση και οχι των ζωων των ζωων και κυριως πρεπει βεβαια να τονωθει η επιτοπου καταναλωση δηλαδη η παραγωγη σφαγη καταναλωση και τελος και η διατάξεις που θα ψηφιστούν πρέπει ε, να κατευθύνονται προς αυτήν την κατεύθυνση. Άλλωστε είναι σημαντικό και για την ανάπτυξη των περιφερειών. Το πρόβλημα που αναφύεται και πάλι και που έχουμε ξανασυζητήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι της μείωσης των χρόνων μεταφορών των ε, ζών των σε 8 ώρες που, μέχρι, που αυτό μάλιστα έχει γίνει και αντικείμενο ε, αναφοράς Ευρωπαίων πολιτών με συλλογή άνω του ενός εκατομμυρίου υπογραφών. Και αυτό πρέπει βέβαια να ε, σημειωθεί επίσης. Προτείνω λοιπόν στο κείμενό μου να πούμε ότι πρέπει να περιληφθεί και αυτό, δηλαδή ο περιορισμός σε 8 ώρες, αυτό βέβαια χρειάζεται περισσότερη συζήτηση, περαιτέρω συζήτηση, αν και θα τεθεί θέμα και εξαιρέσεων όταν υπάρχουν ειδικέ γεωγραφικέ ή άλλες συνθήκες για το αν θα είναι δυνατόν να τηρηθούν τα ωράρια αυτά. Αλλά γενικά ο στόχος θα πρέπει να είναι αυτός. Δηλαδή να αποτελούν μάλλον εξαίρεση οι μεταφορέ που διαρκούν πάνω από 8 ώρες. Το άλλο θέμα είναι το θέμα των ελέγχων των μεταφορών. Η Κομισιόν μας προσφέρει πολλά στοιχεία για τους ελέγχους, ομολογεί όμως η ίδια ότι το σύστημα των ελέγχων δεν είναι ενιαίο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αρμοδιότητες αλλά και η πρακτική ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Το ίδιο ισχύει για, την, για τις επιθεωρήσεις, για το monitoring Υπάρχει και εκεί κάποια πρόοδος, αλλά δεν ε, λειτουργεί πλήρως το σύστημα ελέγχων. Έλεγχοι οι οποίοι πρέπει να ενισχυθούν. Πρόκειται άλλωστε για την πρακτική εφαρμογή εν τέλει των διατάξεων αυτών. Και αυτό δεν αναφέρεται μόναχα στις μεταφορές, αλλά στο σύνολο των διατάξεων προστασίας των ζώων. Η πρότασή μου είναι, εγώ τουλάχιστον αυτό σκοπό να κάνω στην έκθεσή μου, να τονίσουμε δηλαδή ότι στις χώρες μέλη, διότι άλλωστε αυτό εμπίπτει ε, στις αρμοδιότητες των χωρών μελών, στις χώρες μέλη λοιπόν θα πρέπει να δημιουργηθούν εξειδικευμένα όργανα, εξειδικευμένες αρχές που να ασχολούνται με την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Διότι εμείς εδώ ναι μεν εκδίδουμε οδηγίες και κανονισμούς, αλλά όταν εγκύψει κανείς τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στην πράξη, τα συμπεράσματα που διαπιστώνονται είναι ότι είτε η έλεγχη είναι ανεπαρκής, είτε ότι δεν υπάρχουν και καθόλου, δεν αντιδρούν καθόλου τα ελεγκτικά όργανα. Αυτή είναι η εμπειρία πολλών χωρών μελών και της Πολωνίας. Οι οργανισμοί ελέγχου ασχολούνται με την υγεία των ζώων και με την πρακτική εφαρμογή των κανονισμών, αλλά αυτό είναι ένας από τους ε, χώρους ε, Αρμοδιότητά του. Αυτό είναι, ε, αυτό είναι υπόθεση της κτηνιατρικής υπηρεσίας. Βεβαίως εμπλέκεται και η τροχέα για, την τήρηση των χρόνων ε, ε, των διαδρομών κτλ. Άρα είναι κάπως επιφανειακό τελικά το σύστημα ελέγχων και δεν εξασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. το να θεσπιστούν και άλλες διατάξεις για την προστασία των ζώων ενώ δεν τηρούνται οι φυστάμενες θα ήταν υπερβολή. Γι' αυτό εγώ προτείνω να ενισχυθεί το σύστημα ελέγχων, να δημιουργηθούν εξειδικευμένα όργανα, τα οποία δεν χρειάζεται να είναι και μεγάλα, αλλά να είναι όργανα τα οποία κυρίως θα ασχολούνται με τους ελέγχους αυτούς και να μην είναι κατά κάποιο τρόπο παρεργό του αυτό. Αυτά θα είναι, αυτές θα είναι οι κυριότερες πτυχές της εκθεσιό μου. Είμαι πεπισμένος και κατανοώ βέβαια τις ανάγκες των μεταφορών αλλά και τη σημασία των μεταφορών χωρί όμω αυτό να θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο σε μια αγορά που λειτουργεί φυσιολογικά θα έπρεπε να είναι σημαντικό πρόβλημα. Θα πρέπει να φροντίσουμε κυρίως ότι η παραγωγή, εκτροφή δηλαδή, η σφαγή και διάθεση στην εμπορία, στην αγορά, να είναι σε κάπως περιορισμένα γεωγραφικά πλαίσια. Να μην κινούνται τα ζώα ανά την Ευρώπη για να γίνουν όλα αυτά, διότι αυτό ούτε προς το συμφέρον των καταναλωτών είναι, ούτε προς το συμφέρον των ζώων εν τέλει. Και ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσεται στην βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιφερειών. Θα πρέπει να ενισχυθούν ιδιαίτερα τα μικρά σφαγεία και να φροντίσουμε ώστε και η μεταποίηση να γίνεται κοντά στους τόπους εκτροφής των ζώων. Οι δεν μεταφορές. Οι μεταφορές είναι πολύ ευκολότερο να γίνουν εφόσον το αντικείμενο μεταφοράς είναι το κρέας ή τα προϊόντα κρέατος και όχι τα ζωντανά ζώα. Αυτό είναι λοιπόν όπως είπα το βασικό περιεχόμενο της εκθεσιός μου και ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. ευχαριστώ η κυρία Ελισάβετ Γέγκλε. Δεν θα προκαταλάβω τα όσα υποθέτω ότι θα πει η σκιώδη συγκίτριά μας, αλλά θέλω να πω ορισμένα λόγια και αφού πρώτα ευχαριστήσω βέβαια τον εισηγητή που θεωρώ ότι έχει περιλάβει στην έκθεσή του μερικά πολύ σωστά πράγματα και που έχουν πραγματικά και όραμα. Δηλαδή είναι πολύ καλύτερα να μεταφέρεται το κρέας παρά τα ζώντα ζώα. Αυτό είναι από τα πιο σημαντικά επιχειρήματα που έχουμε πλέον πάλι τη δυνατότητα να τα συζητούμε διότι κάποτε ήταν αδύνατον να συζητηθεί το θέμα αυτό. Είχαμε πει τότε ότι ε, τα μικρά σφαγεία δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υγιεινής και επομένως θα έπρεπε να ε, μην ενισχύονται. Θα πρέπει λοιπόν, αφού έχουμε καταλήξει τώρα στο να έχουν περιοριστεί πολύ τα μικρά σφαγεία και να έχουν κυρίως, έχουμε κυρίως μεγάλα και βέβαια συγκεντρωμένα, θα ξαναδούμε τώρα το θέμα, το οποίο είναι βέβαια και προς όφελος της προστασίας των ζώων. Μπορεί αυτό να περιληφθεί και σε διάφορες τροπολογίες, αλλά και το εμπόριο ενδιαφέρεται και οι καταναλωτές. Το εμπόριο έχει δύναμη και μπορεί να επικαλεστεί και το επιχείρημα της προστασίας των ζώων. εγώ το θεωρώ ε, σημαντικό. Από τη Βάρδη, από τη Βάρδη της Γερμανίας που προέρχομαι, είχαμε πει από πάντοτε ότι 8 ώρες έχει καλός. Αλλά σε 8 ώρες πρέπει να περιλαμβάνεται και ο χρόνος φόρτωσης. Τώρα εγώ νομίζω ότι δεν είναι σωστό να πούμε ε, ένα συγκεκριμένο όριο ωρών, ας πούμε για τις κότες 8 ώρες είναι ήδη υπερβολικά μακρόχρονικό διάστημα. Για άλλα ζώα το αντέχουν ευκολότερα. Για πολύ καιρό έχουμε ασχοληθεί υπερβολικά με το χρόνο. Πρέπει να δούμε και τον τρόπο των, ε, της φόρτωσης, της εκφόρτωσης Επίσης η ώρα ανάπαυσης των ζώων ανάμεσα στα δύο τμήματα μεταφοράς αν θα πρέπει να εκφορτωθούν και μετά να ξαναφορτωθούν στο αυτοκίνητο το οποίο πάλι είναι παραγόντας ε, στρες για το ζώο. Είναι λοιπόν πράγματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν. Σε μία ε, εκδήλωση που έγινε χθε, άκουσα ότι η αντιμετώπιση των ζώων, δηλαδή ο τρόπος χειρισμού των ζώων από τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με το καθήκον αυτό και οι γνώσεις των προσώπων αυτών. Και αυτό ήταν ένα θέμα ήδη από το 2005. Τα προβλήματα τα οποία ήδη δεν λύθηκαν με την έκθεση του 2005, ο, ο έλεγχος καθυστερεί, η εφαρμογή, επιβολή βεβαίως των κανόνων αυτών είναι θέμα χωρών μελών και βέβαια οι δυσκολίες πράγματι είναι τέτοιες όπως τις εξήγησε ο εισηγητής. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι έχουμε και διαφορετική ερμηνεία του κανονισμού από τις διάφορες χώρες μέλη. Να, και αυτό λοιπόν πρέπει να συζητηθεί και βέβαια εγώ γνωρίζω από καιρό και δεν ξέρω βέβαια αν ισχύει για όλες τις χώρες μέλη το πρόβλημα των πολλαπλών επιπέδων των ε, φορτηγών αυτοκινήτων που μεταφέρονται τα ζώα. Για παράδειγμα για τα βοηδή είναι διόροφα τα αυτοκίνητα. Όμως τα σημερινά μεταφορικά οχήματα δεν έχουν το απαραίτητο ύψος ώστε τα μεγάλα ε, βοηδή να μπορούν να φορτωθούν και να έχουν κάποιο χώρο πάνω από το κεφάλι τους, δηλαδή ε, συμπιέζονται, δηλαδή ο μεταφορέας βάζει τα ζώα με σε διόροφο, ας πούμε, το εισαγωγικών όχημα, Ωστόσο υπάρχει το πρόβλημα ότι υπάρχει το όριο των 4 μέτρων για τα φορτηγά αυτοκίνητα οι γέφυρε επίση των αυτοκινητοδρόμων δεν είναι παραπάνω από 4 μέτρα πολύ συχνά, άρα πρέπει να μπορούν να περνούν από κάτω τα αυτοκίνητα. Τα φορτώνουν μέσα λοιπόν, μετά κατεβάζουν την οροφή. Και αυτό σημαίνει ότι το ζώο δεν έχει χώρο πάνω από το κεφάλι του. Με αποτέλεσμα έντονο στρες. Αυτά λοιπόν είχα να ε, συνεισφέρω στη συζήτηση. Η κυρία Πόλσεν νομίζω ε, συμφωνεί μαζί μου και συμφωνούμε άλλωστε και για τη στρατηγική την προστασία των ζώων και για την αξιολόγηση των, ε, του θέματος και νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια ευρία προσέγγιση που να περιλαμβάνει και τους αγρότες χωρίς όμως να τους επιβαρύνει επιπροσθέτως οικονομικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό χρειαζόμαστε την συμβολή και του εμπορίου και των καταναλωτών η προστασία των ζώων αφορά όλους. Όλοι άλλωστε ζητούν να τη λάβουμε σοβαρότερα υπόψη. Άρα και όλοι εδώ πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες των. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ κύριε Ισηγητά. Ευχαριστώ για την υποστήριξη που προσφέρατε στον Ισηγητή. Η κυρία Πόλσεν τώρα και μετά Γκάμπαχ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί είναι φιλόδοξο το έργο που έχει αναλάβει να επιτελέσει. Συμφωνώ με αυτό που είπατε για τα σφαγεία. Σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι πρέπει να απαιτήσουμε να γίνει και ένας ε, έλεγχος υγειονομικός. Δεν ήμουν εισηγήτρια, ήμουν σκιώδη εισηγήτρια στην σχετική έκθεση. Αλλά από τη δική μου εμπειρία στην ε, εκλογική μου περιφέρεια μπορώ να σας πω ότι οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, στη Βορειοσουηδία δηλαδή. Τεράστιες αποστάσεις διανύονται. Πώς θα έχουμε εξορθολογισμό της κατάστασης με τα σφαγεία. Πώς είναι δυνατόν τα ζώα να μπορέσουν να αντέξουν ε, μία δωδεκάωρη και πάνω μεταφορά μέχρι το σφαγείο. Δεν είναι δυνατόν. Και σε ό,τι αφορά το δεύτερο πυλώνα, για τις περιφέρειες συγκεκριμένα. Και όχι τόσο τις μεταφορές, αλλά πρέπει να σας πω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό που προτείνει είναι κάποιες κατευθύνσεις, guidelines. Και αυτό πραγματικά με ξενίζει. Διότι απ' την άλλη, σύμφωνα με τον οργανισμό EFSA για την ασφάλεια των τροφίμων, βλέπουμε να υπάρχει κάποια διαφορά σε σχέση με τα επιστημονικά στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Δηλαδή, επί της ουσίας, δεν σεβόμαστε μια βασική αρχή. Ότι δηλαδή θα πρέπει η δική μας νομοθεσία να βασίζεται στα επιστημονικά στοιχεία. Κάτι που δεν συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση και αυτό για μένα είναι πολύ σοβαρό. Άρα θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός αυτός, ώστε να γίνονται σεβαστά τα επιστημονικά στοιχεία, επιστημονικές αποδείξεις. Θέλουμε οι πολίτες να είναι πιο κοντά σε εμά και θέλουμε ίσως και να καταλάβουν στην προκειμένη περίπτωση τι συνεπάγεται η πολύωρη μεταφορά των ζώων. Μπορούμε όμως στην νομοθεσία να επιβάλλουμε μια προθεσμία των 8 ωρών. Δεν είμαι σίγουρη γιατί για ε, τη μεταφορά των ζώων και υπό συγκεκριμένε συνθήκε, οι επιστήμονε λένε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένα είδη ζώων, για συγκεκριμένα ζώα. Άλλα ζώα και υπό άλλε συνθήκε, ναι, είναι δυνατή και μια ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια ενδεχομένως μεταφοράς τους. Είναι λίγο αόριστα τα πράγματα. Είναι λίγο ασαφής η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Εμείς είμαστε στη μέση. Απ' τη μια είναι οι πολίτες και από την άλλη οι επιστήμονες. Και εμείς στη μέση. Άρα πρέπει να το σκεφτούμε δύο και τρεις φορές πριν προτείνουμε τη λύση για το μέλλον. Γιατί πρέπει να βρούμε μια λύση καλή για τα ζώα, αλλά και για την οικονομία, αλλά και για την κοινωνία. Υποθέτω ότι η καλύτερη οικονομική λύση είναι να ξαναδημιουργήσουμε περιφερειακά σφαγεία, τοπικά σφαγεία αφού θέλουμε να μεταφέρουμε κρέας και όχι ζώντα ζώα. Εάν θέλουμε να μεταφέρουμε κρέας όμως, αυτό το κρέας πρέπει ουσιαστικά να είναι μεταποιημένο. Ακόμη και τα σφάγια να τα μεταφέρουμε, αυτό είναι πιο αποτελεσματικό από το να μεταφέρουμε ζώντα ζώα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή και νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε ένα δύσκολο πρόβλημα μεταξύ άλλων και διότι προσπαθούμε με κανονισμούς να διορθώσουμε πράγματα τα οποία ε, διαρθρωτικά είναι πλέον εσφαλμένα. Ο κανονισμός κυρίως ασχολείται με την προστασία των ζώων και με τις μακρινές διαδρομές. Το πρόβλημα όμως είναι και το πώς έχουμε διαμορφώσει τη γεωργία μας στην Ευρώπη. Δηλαδή κάτι που κατά τη γνώμη μου πρέπει να μας απασχολεί πάντοτε. Δηλαδή, μόνο με τον παρόντα κανονισμό δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση ούτε της εκτροφής των ζώων, της εκτροφίας ε, συνολικότερα, ούτε και της μεταποίησης του προϊόντος. Θα χρειαστούμε μια διαφορετική γεωργία. Θα συμφωνήσω με την κυρία Πόλσεν ότι 8 ώρες είναι συμβολικές για την κατάσταση. Δηλαδή, έχουμε στην Ευρώπη μια κατάσταση όπου τα ζώα λόγω του τρόπου που μεταφέρονται στην ουσία δεχόμαστε εμείς ότι θα πάσχουν τα ζώα. Από την άλλη μεριά υπάρχουν περιοχές στην Ευρώπη που καταναλώνουν περισσότερο κρέας από ό,τι παράγεται, από αυτό που παράγεται τοπικά. Άρα και θα χρειαστεί μεταφορά. Βέβαια, η μεταφορά να είναι μεταφορά κρέατος και όχι μεταφορά ζωντανού ζώου. Αυτό που αποσκοπούμε τώρα είναι να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όπως είναι τώρα. Και από αυτά που λέει η ΕΦΣΑ, τίθεται και το ερώτημα πώς μπορούν να μεταφέρονται τα ζώα σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε είδου. Θα θυμίσω ε, ένα από τα συμπεράσματα του κυρίου Σλούτερ Φανταστείτε διαστάσεις ενός διπλού κρεβατιού και πάνω σε αυτό να μεταφέρονται τέσσερις αγελάδες ή δέκα πρόβατα. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες να είναι και διαφορετικά τα πράγματα. Και διορωτώ με αν αυτό μπορεί να γίνει σε, στα πλαίσια άλλων δομών, για παράδειγμα, μέσα στην προσπάθεια ανάπτυξη τη υπαίθρου. Να δημιουργηθούν δομέ δηλαδή, οι οποίε να επιτρέψουν συντομότερες διαδρομέ. Εμείς έχουμε βέβαια καταθέσει ορισμένε τροπολογίε με τι οποίε δεν έχουμε συμφωνήσει, για τι οποίε μάλλον δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμη με τον ε, εισηγητή, αλλά που νομίζουμε ότι είναι προ την σωστή κατεύθυνση, δηλαδή οι μεταφορέ να γίνονται σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα τη επιστήμη, σε άλλου τομεί να δημιουργηθούν οι προποθέσει, όπω άλλωστε συζητήθηκε σήμερα, για παράδειγμα τα περιφερειακά ή τοπικά σφαγεία. Αυτά βέβαια είναι όλα χρήσιμα. Νομίζω όμω ότι για την ώρα δεν πρέπει να χάσουμε, να πετάξουμε όπως λένε και το μωρό μαζί με το νερό του, του λούτρου, αλλά να μην λησμονούμε ότι δεν μπορούμε να δούμε μονάχα τώρα την κρίση η οποία όντως επιβάλλει ορισμένα πράγματα και να λησμονήσουμε τελείως την προστασία των ζώων. Αυτό που θεωρώ πάντως ότι χρειαζόμαστε στο μέλλον είναι μια διαφορετική γεωργική πολιτική. Ευχαριστώ. Κυρία Μαγκίνες. Και μετά Ντερ Λάγκ ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν με θέλουν τα μικρόφωνα σήμερα. Πολύ σύντομα. Υποστήριζω την άποψη της κυρίας Πόλσεν για επιστημονική τεκμηρίωση Υπάρχει κίνδυνος όταν ε, λαμβάνουμε υπόψη το χρόνο μεταφοράς. Ε, μπορούμε να έχουμε ε, πολύ κακές συνθήκες ακόμα και μέσα σε μισή ώρα και μπορεί τα ζώα να ταξιδεύουν πολύ πιο άνετα ακόμα και να ταξιδεύουν επί 16 συναπτές ώρες. Συναπτές ώρες. Ε, Επομένω, πρέπει να κάνουμε υπόψη μας τα επιστημονικά στοιχεία που έχουμε για το χρόνο μεταφοράς. Η έκθεση της Κομισιόν ήταν πολύ χρήσιμη, γιατί μας είπε τι πέτυχε ο κανονισμός. Υπάρχει και ένα πρόβλημα εφαρμογή βέβαια του κανονισμού. Ε, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα έλλειψη εφαρμογή ε, στην πραγματικότητα ψάχνουμε να νομοθετήσουμε περαιτέρω, αντί να εφαρμόσουμε αυτά που ήδη έχουμε. Ε, η ανησυχία μου λοιπόν είναι αυτή. Α δούμε τι έχουμε και α προσπαθήσουμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη να τα εφαρμόσουν όλα όσα έχουμε. Η κυρία Γέγκλε ε, έκανε κάποια σχόλια χρήσιμα. Μίλησε για τη δική τη ε, περίπτωση, τη δική τη κατάσταση, για τη σφαγή και τα σφαγεία. Και ότι σε ορισμένε περιοχές Ευρώπης υπάρχουν κάποια προβλήματα. Ας δούμε λοιπόν όμως το εμπόριο στην Ευρώπη γενικά. Εμείς μεταφέρουμε νεότερα ζώα. Αν δείτε τι επενδύσει και την έκθεση της Κομισιόν που αναγνωρίζει ότι έχει γίνει, τι έχει γίνει από τις εταιρείε μεταφοράς, έχουν δηλαδή αγοράσει εξειδικευμένα οχήματα, ώστε να φροντίζουμε τα ζώα και να τα αντιμετωπίζουμε καλά. Ε, υπάρχει κατάρτιση. Ε, πρέπει να δούμε τις καλές πρακτικές, τις βέλτιστες πρακτικές στο τομέα αυτό και να προσπαθήσουμε να πείσουμε και τους υπόλοιπους να αυξήσουν τα πρότυπα. Ε, μιλήσατε για ένα νέο εξειδικευμένο φορέα, κύριε Σιγητά, μπορείτε να το, θα μπορούσατε να το σχολιάσετε περαιτέρω. Όπω είπε και ένα άλλο συνάδελφο, θα πρέπει να μην ξεχνάμε και τα προγράμματα λιτότητα στην Ευρώπη και ότι δυσκολεύονται οι δημόσιοι φορεί να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα σε τέτοια θέματα. Πώς μπορούμε να πετύχουμε τις ε, βέλτιστες πρακτικές χωρίς να αυξήσουμε υπερβολικά το κόστος. Η μεταφορά των ζώων των ζώων είναι ε, εγγενές στοιχείο της ε, Ιρλανδικής κτηνοτροφίας. Έχουμε κάνει επενδύσεις ούτως ώστε να γίνονται μεταφορές χωρίς να ξεχνάμε την ευμερία των ζώων. Αυτό είναι κλειδί, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι κανονισμοί που έχουμε εφαρμόζονται σωστά. Αντί να μειώνουμε απλώς τους χρόνους ε, μεταφοράς χωρίς να βελτιώνουμε στην πραγματικότητα καθόλου ούτε στο παραμικρό την ευημερία των ζώων. Ευχαριστώ. Κύριε Ντελάγκα. Και μετά Γκαρσία Περές. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεση. Νόμιζα ότι είναι πολύ συναισθηματικά φορτισμένο. Είναι συναισθηματικά φορτισμένο το θέμα. Και ακούγονται πολύ διαφορετικές απόψεις. Για την ε, ομάδα μου αυτό που είναι σημαντικότερο από όλα είναι ότι αυτή η έκθεση είναι ισορροπημένη. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία θέματα. Καταρχάς, ένα θέμα που έθεσε και η κυρία Μαγκίνης. Δηλαδή, όντως θα πρέπει να εστιάσουμε ε, σε αυτούς που δεν εφαρμόζουν τους κανόνες. Υπάρχουν όμως και πολλοί μεταφορείς που παρά τη, τους χαλεπούς οικονομικούς καιρούς έκαναν σημαντικές επενδύσεις, αγόρασαν νέα οχήματα, ε, σε προγράμματα, έκαναν επενδύσεις σε προγράμματα κατάρτισης. Ε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και ότι πολλά πράγματα πηγαίνουν καλά, όχι μόνο στραβά. Επίσης υπάρχει θέμα με τους ελέγχους στα κράτη-μέλη. Αλλά τώρα μοιάζει να αντιμετωπίζουμε όλα τα κράτη-μέλη με τον ίδιο τρόπο. Ότι όλα τα κράτη-μέλη είναι κάκιστα. Ε, δεν έχουν αποτελεσματικούς ελέγχους. Και αν δείτε τη μεταφορά των ε, ζώων σε όλη την Ευρώπη, βλέπετε ότι η διάφορα κράτη-μέλη είναι πιο αυστηρά από κάποια άλλα. Υπάρχουν καλοί και κακοί ελεγχτές παντού. Αν δείτε ε, μεταφορές ε, ζώων που παρακάμπτουν κάποιες χώρες, τότε τι, είναι το συμπέρασμα, ότι η συγκεκριμένη χώρα είναι πιο αυστηρή από τη γειτονική. Τι θα κάνουμε με αυτό. Τι θα κάνουμε με το γεγονός ότι ε, κυρώσεις και πρόστιμα είναι τόσο διαφορετικά που μπορεί να πληρώσεις ας πούμε σε ένα κρατός 50 και σε ένα άλλο μερικές χιλιάδες ευρώ. Δεν έχουμε την αρμοδιότητα εμείς να καθορίσουμε τα πρόστιμα, αλλά θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο φιλόδοξοι από τη σημερινή κατάσταση που αφήνουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν ό,τι ακριβώς θέλουν. Εντάξει. Μην ξεχνάμε λοιπόν όμως ότι κάποια κράτη-μέλη είναι αυστηρότερα και από τα άλλα για τη διάρκεια του ταξιδιού μεταφοράς. Ε, αν δεν προσέξουμε, η έκθεση αυτή θα μιλάει μόνο για τις 8 ώρες. Αν τελικά είναι μια τέτοια έκθεση, ε, δεν νομίζω ότι θα εξασφαλίσει η ευρεία πλειοψηφία, ούτε καν πλειοψηφία, αν μιλάει μόνο για το χρόνο μεταφοράς. Ε, αυτή τη στιγμή κυρίως γι' αυτό μιλάει. Ιδανικά δεν θα πρέπει να εστιάζουμε στο χρόνο ε, μεταφοράς, αλλά στι συνθήκες μεταφοράς. Το μόνο πρόβλημα είναι, είναι ότι στην περίπτωση της φαγής ειδικά, ε, εκεί έχουμε τα περισσότερα προβλήματα κατά τη μεταφορά, όταν ε, στο τέλος είναι, ακολουθεί η σφαγή. Γι' αυτό μην ξεχνάμε την έκθεση που υιοθετήσαμε εμεί ω Κοινοβούλιο το 2004 και να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στα ζώα προσφαγή, γιατί όντω θα πρέπει να προωθήσουμε τη, σφα... τη σφαγή στην περιοχή, να βάλουμε ε, ως όριο τις 8 ώρες και να κάνουμε μια μικρή εξαίρεση για την Ιρλανδία, αλλά για τα ζώα προσφαγή να πούμε 8 ώρες, αλλά για τα ζώα προς εκτροφή ή προσπάχυνση που έχουν πολύ υψηλότερη αξία στο τέλος της μεταφοράς να εστιάσουμε στις συνθήκες. Νομίζω ότι το 2004 φτιάξαμε μια ωραία έκθεση. Η κυρία Γιάγκλε είπε όχι μόνο να έχουμε τους γεωργούς αλλά και τους μεταφορείς και τους καταναλωτές και τους ακτιβιστές υπέρ της ευημερίας των ζώων ε, πίσω μας και υπέρ της έκθεσής μας. Το 2004 τους είχαμε τους αυτούς μαζί μας με την έκθεσή μας. Α την κρατήσουμε λοιπόν αυτή τη 2004 και αμαγκίνες τώρα. Εν μέρη είναι νέα νομοθεσία όντω. Αλλά από την άλλη καλό θα ήταν να στείλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Συμβούλιο ε, αυτό το μήνυμα. Να πει, κοιτάξτε, πριν από 10 χρόνια εμεί αυτό προτείναμε. Ε, και επειδή τότε δεν είχαμε τη συναπόφαση, εσεί αποφασίσατε τότε να μα αγνοήσετε εντελώ και να εστιάσετε μόνο στι συνθήκε μεταφορά. Το να εστιάσετε στι συνθήκε μεταφορά και μόνο με την ε, αδυναμία που έχουμε να επιβάλλουμε σωστούς ελέγχους, δεν θα λειτουργήσει ποτέ. Ας είμαστε λοιπόν ρεαλιστές. Λοιπόν, επομένως, για τα ζώα προσφαγή μιλήστε για 8 άωρο, αλλά για τα υπόλοιπα ζώα να λάβουμε υπόψη μας τα στοιχεία και να λάβουμε υπόψη και τις συνθήκες μεταφορές, μεταφοράς. Ε, έχουμε αυτή την απαρχή που είναι η έκθεση του εισηγητή. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Ε, το ΕΛΤ θα κάνει και προτάσεις, ούτως ώστε να εξισορροπηθεί περισσότερο η έκθεση. Είμαι διατεθειμένη να συνεργαστώ με τους υπόλοιπους σκιώδεις εισηγητές για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Είναι τρομακτικό να το λέω αυτό στην ηλικία που έχω φτάσει, αλλά ας εμπνευστούμε από την έκθεση που φτιάξαμε πριν από 10 χρόνια. Μια χαρά ήταν. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκαρσία Περές. Και μετά ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή ο οποίος μας παρουσίασε το σχέδιο έκθεσης. Μπορώ να πω ότι συμφωνώ εν γέννη με την έκθεση, με τις αρχές, δηλαδή της καλής μεταχείρισης των ζώων, τους όρους μεταφοράς και ούτω καθεξής. Παρ' όλα αυτά θέλω να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένη σε κάποια θέματα τα οποία έθεσαν και ορισμένοι από τους προλαλήσαντες συναδέλφους μου στην διάρκεια της συζήτησης. Θεωρώ ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής είναι ισορροπημένη, εκείνη από τη βάση ότι η ρυθμίσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι οι κατάλληλες. Να μην δημιουργήσουμε λοιπόν νέες ρυθμίσεις, όπως λέγει η κυρία Μαγκίνες. Σημαντικό είναι να εγγυηθούμε την εφαρμογή, την πρακτική εφαρμογή των ρυθμίσεων που έχουμε ήδη αυτή τη στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν καθορίζει κάποιες δράσεις ε, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν τοπιστεί και για να είναι ε, καλύτερη εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων ρυθμίσεων. Συμφωνώ απόλυτα. Η μεταφορά των ζώων είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για οικονομικούς λόγους. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια μεγαλύτερη οικονομική αξία στον τόπο ε, προορισμού και οι φορείς εκμετάλλευσης είναι αυτοί που έχουν ε, και το μεγαλύτερο όφελος από τη βελτίωση της όλης κατάστασης. Αν όμω ε, αυτό το οποίο μα απασχολεί είναι και η καλή μεταχείριση των ζώων στη διάρκεια τη μεταφορά του, αυτό ο στόχο θα πρέπει να επιδιώκεται ε, σε όλη την διάρκεια, σε όλη μάλλον τη μεταφορά ε, των ζώων. Όχι μόνο για τη μεταφορά των ζώων που προορίζονται προ φαγή. Συμφωνώ με κάτι που είπε η κυρία Πάουλσεν και επανέλαβαν και άλλοι συνάδελφοι σε σχέση με το ότι οποιοδήποτε μέτρο αυτό θα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία για κάθε ζώο συγκεκριμένα. Αυτό το οχτάωρο δεν έχει κάποια επιστημονική βάση. Η ΕΦΣΑ για τη μεταφορά χείρων λέει ότι το στρες που βιώνουν τα ζώα είναι το ίδιο, ανεξαρτήτως της διάρκειας. Ένα άλλο παράδειγμα. Αυτό που είναι καλό για τα, ζώα, για τα υποειδή, ε, τα άλογα, ότι θα πρέπει να σταματούν, να τα ξεφορτώνουν και να τα ε, βάζουν λίγο να περπατήσουν, αυτό είναι αντιπαραγωγικό για άλλα ζώα, άλλα είδη ζώων. Επομένως πάλι δεν πρέπει να εφαρμοστεί αδιακρίτως. Επίσης, μιλάμε για ευρωπαϊκό ε, νομοθέτημα, άρα δεν πρέπει να ξεχνάμε τις γενικές αρχές. Όταν θέλουμε να δρομολογήσουμε ενδιαφέροντα και κατάλληλα μέτρα. Η Επιτροπή μας πρέπει να έχει επίγνωση και με βέβαια ότι ισχύει αυτό. Ε, πρέπει να έχει υπόψη τι επιπτώσει που θα μπορούσαν να υπάρχουν για τη δική μου χώρα, την Ισπανία και για άλλε χώρε ε, που είναι στην περιφέρεια τη Ένωση και που είναι πολύ σημαντική μεταφορά των ζώων και λόγω τη γεωγραφική μα θέση και λόγω των σημαντικών εμπορικών ροών. Η ε, κίνηση δηλαδή ζωντανών ζώων από τη χώρα μα προ άλλα κράτη-μέλη. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι πιστεύω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και αυτή η παράμετρος όταν θα τοποθετηθεί η Επιτροπή Γεωργίας. Είμαι βέβαιο ότι και στη διάρκεια της συζήτησης αλλά και στο πλαίσιο των, της εργασίας που θα πρέπει να γίνει μεταξύ των εισηγητών, σκιωδών και άλλων συναδέλφων θα καταλήξουμε σε μία πρόταση ισορροπημένη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Σάκνιου μετά Χόισλινγκ. Υποστηρίζω όλα όσα είπε η κυρία Μαγκίνες. Και επιπλέον υπάρχει και ένας ηθικό εκβιασμό των πολιτικών, ότι αν ε, φέρουμε αντίρρηση σε οτιδήποτε απαιτεί περισσότερη νομοθεσία, τότε ε, είσαι σκληρός και κακός. Ε, απλώς θα πρέπει να είμαστε λογικοί. Στο Ηνωμένο Βασίλειο Ίσως είμαστε μοναδικοί. Έχουμε το εμπόριο αυτό των ε, προβάτων. Ε, πολλά από τα πρόβατα αυτά ε, γεννιόνται το καλοκαίρι στη βόρειο ε, Σκοτία, αλλά μετά τα, τον υπόλοιπο χρόνο θα πρέπει να τα μεταφέρουμε και χρειάζονται περισσότερο από 8, 8 ώρες για να τα μεταφέρουμε αυτά τα ζώα. Ε, και μην ξεχνάτε ότι δεν μιλάμε για αυτοκινητόδρομους, αλλά για πολύ στενούς ε, ε, δρόμους, οι οποίοι έχουν όλο καμπύλες και τα λοιπά και τα, τα ταξιδεύεις το, πολύ με 30 χιλιόμετρα την ώρα. Άρα δεν φτάνω 8 ώρες, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει ο οδηγός. Ε, εδώ ο εισηγητής μιλάει για ειδικά μέτρα. Να, ορίστε τα ειδικά μέτρα. Η κυρία Γέγκλε μίλησε για τη μεταφορά ορνήθων ε, αυτό το κάνουμε το βράδυ, γιατί τότε κοιμούνται. Ή μάλλον μέσα στο σκοτάδι, συγγνώμη. Γιατί απλώ κοιμούνται και τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για να τι μεταφέρουμε. Ε, Επίση, το φόρτωμα και το ξεφόρτωμα είναι πάρα πολύ. αυξάνει το άγχο, α πούμε. Και αν ο οδηγό οδηγεί έτσι με έναν σταθερό ρυθμό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι στρεσάρονται τα ζώα. Ε, το, το πιο δύσκολο θα ήταν για τα ζώα να τα φορτώνουμε, να τα ξεφορτώνουμε κάθε τρει και λίγο. Επίση, ε, μιλήσατε για περιορισμένε αγορέ, δηλαδή να τα πουλάμε να τα πουλάμε σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό είναι συνταγή για μονοπόλιο. Ε, θα πρέπει να πάνε σε αυτό το σφαγείο, ας πούμε. Ε, δεν μπορούμε να τα στείλουμε πουθενά αλλού. Επίσης, ε, μιλήσατε για τους πολλού ορόφους. Αυτό το χρησιμοποιήσαμε τα του 80. Τότε. Ε, ας πούμε για τα βοηδή, ας πούμε είχαμε δύο α, ορόφους, ε, άλλα, για άλλα ζώα είχαμε τέσσερις ορόφους κτλ. Μπορούσαμε να περάσουμε αυτά τα φορτηγά κάτω από τις ε, γέφυρε. δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Επίσης τα ε, μερικαστικά ταξιδεύουν καλύτερα όταν δεν έχουν φάει. Ναι, εμείς λέμε ότι πρέπει να τα ταΐζουμε, να τα ποτίζουμε και τα λοιπά κατά, κατά το ταξίδι, αλλά τότε μπαίνουν στη διαδικασία μερικασμού. Και φανταστείτε, μένουν εκεί στο φορτηγό, φανταστείτε τη βρώμα. Φανταστείτε. Εγώ νομίζω ότι καλύτερα να τα μεταφέρουμε, ας πούμε, ε, χωρίς φαγητό, ε, κατεβαίνουμε, τα κατεβάζουμε από τη σκοτία, ας πούμε, και τη στιγμή που κατεβαίνουν από το φορτηγό, ε, ωραία και καλά μπορούν να φάνε. Ε, δεν χρειάζεται να τα ταΐζουμε με χρησκασμού. Νομίζω ότι είναι ε, κλιματικό. Γιατί απλώς αν έχουν φάει με σκασμού θα πέσουν ας πούμε, πάνω σε άλλα ζώα, θα ποδοπατηθούν εκεί πέρα, δεν είναι σωστό. Επίσης, ε, δεν είναι σωστό να βάζουμε μεγάλα με μικρά ζώα μαζί, ας πούμε, α, χωρίς χωρίσματα. Ε, επίσης, Υπάρχουν και, τα, και το θέμα των, υπάρχει και το θέμα των κεράτων. Ε, πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας κάτι μεταφορά. Επίσης, ε, έχουμε καμιά φορά ε, έγκυα ζώα ε, που γεννάνε μέσα στα ταξίδια, στο καδιάρι του ταξιδιού. Μην το κάνετε αυτό, μην φορτώνετε έγκυα ζώα. όλα αυτά είναι θέμα κοινή λογικής σε μεγάλο βαθμό. Ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε τώρα τον κύριο Χόισλινγκ. Ασφαλώς και χρειάζεται ανάληψη δράσης, όχι μόνο επειδή το ζητούν ένα εκατομμύριο πολίτες όπως ε, λέχθη προηγουμένως, αλλά και διότι ε, αυξάνονται διαρκώς οι μεταφορές, όπως είπε και ο εισηγητής, άρα έχουν υπάρξει εδώ κάποιες σημαντικές παραλήψεις. Μία από τις αιτίε που οφείλουμε να στιγματίσουμε και την οποία έχουμε προκαλέσει και εμείς βέβαια εν μέρη, διότι κλείσαμε ή οδηγήσαμε στο κλείσιμο πολλά μικρά ε, σφαγεία λόγω των προδιαγραφών υγιεινής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά εδώ πρέπει να γίνει μια διόρθωση και να δούμε και πού το παρακάναμε, πού πρέπει να κάνουμε όπως είπα κάποιες διορθώσεις και να τα αποκαταστήσουμε αυτά και με τις ε, διαρθρώσεις για την ανάπτυξη της υπέρθρου. Βέβαια Υπάρχουν και άλλες αιτίε σχετικές με την προστασία των ζώων, με τη μεταφορά των ζώων, που δεν έχουν σχέση με αυτά, αλλά έχουν σχέση με τις τιμέ. Στη Γερμανία μεταφέρονται πολλά χοιρινά από το βορρά της Γερμανίας στο νότο, γιατί είναι καλύτερες οι τιμέ εκεί. Είναι όμως εντελώς περιττή στην πραγματικότητα η μεταφορά αυτή. Πρέπει λοιπόν να δούμε εάν περιφερειακά μπορεί να γίνει μια ρύθμιση ώστε να μεταφέρεται καλύτερα το κρέας του ζώου παρά το ίδιο του ζώου. Βέβαια αυτό δεν είναι μονάχα ε, το θέμα ορίου, οκταόρου δηλαδή. Οφείλουμε να δούμε ότι οκτάωρο για πολλά ζώα είναι ήδη υπερβολικά μακρά περίοδος και είναι βέβαια και οι συνθήκες της μεταφοράς πάρα πολύ κεντρική σημασία. Είναι λοιπόν ε, εύκολο να πούμε «Α, εντάξει, προσανατολιζόμαστε στο οκτάωρο». Όμως το ζήτημα είναι και πώς διαμορφώνονται οι συνθήκες της μεταφοράς ε, στην πράξη. Λέχθηκε πολλές φορές ότι υπάρχουν ιδιαίτερες δυσχέρειες σε ορισμένες περιφέρειες. Οι περιφέρειες της Βόρειας Ευρώπης, για παράδειγμα, όπου δεν υπάρχει υποδομή για την σφαγή, πρέπει να κάνουμε εξαιρέσεις και για ορισμένα ε, ζώα, όπως για παράδειγμα για άλογα τα οποία συμμετέχουν σε υπηκούς αγώνες, διότι αν δεν επιτρέπουμε τη μεταφορά, πολλοί ε, που τους αρέσουν οι υπηκοί αγώνες δεν θα μπορούν να μεταφέρουν τα άλογά τους. Αυτές οι εξαιρέσεις βέβαια πρέπει να είναι περιορισμένες. Έτσι λοιπόν εκφράζω την ελπίδα και την ευχή ε, με κοινή συνεργασία να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ορθή βάση και να δείξουμε ότι όντως εγκύπτουμε με φροντίδα στο θέμα και αυτό είναι σημαντικό για να γίνει αποδεκτή η λύση που θα προτείνουμε και από τον αγροτικό κόσμο και να δώσουμε απαντήσεις βέβαια και στις ανησυχίες της κοινή γνώμη. Ευχαριστώ κύριε κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι από την ομάδα ECR που είναι και ο εισηγητής και θέλω να τον ευχαριστήσω για το έργο του πάνω σε αυτό το θέμα, που είναι ένα θέμα που μας συγκινεί. Πολλές φορές δεχόμαστε email και πραγματικά είναι ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Πολύ σωστά είπε ο εισηγητής μας ότι πρέπει να υπάρξουν περισσότεροι έλεγχοι ε, των οχημάτων που μεταφέρουν ζώα, για να δούμε πώς μεταφέρονται και με ποιο τρόπο τα μεταχειρίζονται αυτοί οι οποίοι έχουν αναλάβει τη μεταφορά τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, καταρχήν συμφωνώ απόλυτα με το ότι καλό είναι να έχουν σφαγιαστεί τα ζώα στο δυνατόν πιο κοντά ε, στη γεωργική εκμετάλλευση όπου έχουν εκτραφεί. Στη δική μου περιοχή, τα δυτικά Midlands, ε, τα μικρά σφαγεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Και αυτό λόγω εν μέρη και των κανονισμών που ισχύουν στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και που επηρεάζουν τα σφαγεία. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή να μην επιβάλλουμε με καλή πίστη κανονισμού, αλλά τελικά ε, να βλέπουμε αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκαμε. Και τελικά τα ζώα πρέπει να μεταφερθούν πολύ μακρύτερα για τη σφαγή. Με ανησυχεί επίσης το ότι σε, κάποιους, ε, σε κάποιες περιοχές, ιδίως βόρεια, στα βόρεια, ε, στα νησιά Σέτλαντ, για παράδειγμα, στη, στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν μπορούμε. Είναι αδύνατο να εκτρέ, εκτρέφουμε ζώα δεν μπορεί να μεταφερθούν για διάστημα μεγαλύτερο των οκτών, γιατί δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να τα περάσουμε από τα Σέτλαντ στην υπηρετική χώρα. Από ό,τι λέτε εσείς φαίνεται θα υπάρξουν αποκλήσεις, ε, παρεκκλήσεις μάλλον και εξαιρέσεις. Να συμφωνήσω και με τους ε, ορισμένους από τους προλαλήσαντες που είπαν ότι ίσως το βασικό θέμα δεν είναι τόσο ο χρόνος, η διάρκεια της μεταφοράς, αλλά οι συνθήκες της μεταφοράς. Και ανάλογα με το είδος του ζώου μπορεί να διαφέρουν και ανάγκες. Στη δική μου χώρα τα άλογα που στέλνονται προς ε, σφαγή είναι ένα θέμα πολύ συναισθηματικά φορτισμένο. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όταν νομοθετούμε μήπως ε, με το νέο νομοθέτημα δεν πετύχουμε το στόχο που επιδιώκουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γιάρ και μετά Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συζητούμε σήμερα ένα θέμα συναισθηματικά φορτισμένο όπου συχνά έτσι προβάλλονται και εικόνες η μεγάλη κατακραυγή ήταν όταν γίνονταν και πολλές επιδοτήσεις εξαγωγών και μεταφέρονταν τότε ζώα σε όλες τις γωνιές της Ευρώπης και οι εικόνες ήταν όντως τρομακτικές. Είχα συνομιλήσει με ένα μεταφορέα τότε, off the record όπως λένε, και μιλώ βέβαια και για μια περίοδο όπου υπήρχαν και δυσχέρειες της διαβάσης των συνόρων κτλ. Και ήταν πραγματικά απαράδεκτα τα πράγματα αυτά. Αυτές οι εικόνες όμως ακόμα έχουν μείνει στη, στο νου της κοινή γνώμη και αυτά θυμάται όταν ε, μιλούμε για μεταφορές ζώων. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ ευαίσθητοι αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστές. Έχω σημειώσει βέβαια ορισμένα πράγματα και μία από τις φράσεις που έχω ε, σημειώσει είναι ότι πρέπει να βασιστούμε στην έκθεση που είχε ψηφιστεί εδώ προ δεκαετίας εγώ βέβαια δεν ήμουν τότε εδώ παρόν. Ναι, ναι, ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία κύριε Γέγκρε, καλά το είπατε. Η έκθεση δεν ήταν άσχημη βέβαια. Εφόσον κάνουμε, εφόσον συντάσσουμε έκθεση τώρα και έχουμε την δυνατότητα να συμμετάσχουν και οι χωρισμένοι, διότι δεν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, διότι και να αποφασίζουμε εδώ στην Ευρώπη και εγκρίνουμε, εφόσον δεν εφαρμόζονται, οι κακές, οι τρομακτικές εικόνες θα μας ξανάρθουν πίσω να μας κυνηγούν και ο καταναλωτής αντιδρά εξοργισμένος. Ωραία, απλή λύση είναι το 8 Όμως έχουμε μεγάλη ευθύνη και συμφωνώ και με τους υπολείπους ότι υπάρχει διασύνδεσμος μεταξύ του είδους του ζωού, της μεταφοράς, ε, του, του χρόνου μεταφοράς και των συνθήκων. Το ίδιο και ένας άνθρωπος άλλο, άλλο ε, ε, μια διαδρομή μιας ώρας σε ένα αστικό λεωφορείο και άλλο 20 ωρών σε ένα αναπαυτικό πούλμαν που πηγαίνει μακριά. Τα είπαμε αυτά βέβαια, τα είπαν και άλλοι συναδελφοί. Πρέπει να φροντίσουμε και διαρθρωτικά να μειωθούν οι μακρινές μεταφορές, τοπικά και περιφερειακά σφαγεία ήδη και καταφέραμε όντως και εμείς στο Όντενβουρκ να έχουμε κρεοπολία τα οποία παλαιότερα μάλιστα είχαν την έγκριση να προβαίνουν στη σφαγή και οι ίδιοι. Φροντίσαμε τώρα με τις προδιαγραφές υγιεινής να μην τους, ε, να μην τους επιτρέπεται. Και καταλήγουμε στην ανοησία να πρέπει να πρέπει τα ζώα που παράγονται επί τόπου σε εμά, εκεί όπου υπάρχουν και τα κρεοπολία, να πρέπει πρώτα να μεταφερθούν 50 χιλιόμετρα μακριά στο σφαγείο και μετά να επιστρέψουν τα σφάγια στους κρεοπόλες. Άρα να επαναφέρουμε τα μικρά ε, ε, σφαγεία, να δοθεί και η δυνατότητα σφαγής ευρύτερα, με βέβαια ε, σωστά τηρούμενες προδιαγραφές υγιεινής. Dziękuję, Νομίζω ότι τελειώσαμε εδώ με τον κατάλογο μιλητών και μπορούμε να ακούσουμε τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα. Νομίζω ότι η συζήτηση ήταν ε, πάρα πολύ διεξοδική όλες οι πτυχές της έκθεσης νομίζω καλύφθηκαν από τους βουλευτές, πόσο πολύπλοκο είναι να καθορίσουμε τη διάρκεια της μεταφοράς, πόσο δύσκολο κάποιες φορές είναι να συμφιλειωθούν οι επιστημονικές απόψεις με τα κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει ε, και από την έκθεση της, Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ο βασικός μας στόχος είναι να ενισχύσουμε την εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων. Για να συμπληρώσω τις πολύ αναλυτικές και εμπεριστατωμένες παρεμβάσει. να πω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονό ότι οι ότι ο κοινωνικο-οικονομικός κόσμος εξελίσσεται. Αφού αυτού έχουμε ιδιωτικέ πρωτοβουλίες, πάρα πολύ θετικέ. σε ό,τι αφορά τις καλές πρακτικές, για παράδειγμα, και βέβαια χρειάζεται χρόνο. Μιλήσαμε και για την εκπαίδευση. Ο κανονισμό ε, εγκρίθηκε το 5, αλλά τέθηκε σε ισχύ το 7. Έχουμε δηλαδή πλέον ε, κάποια χρόνια ε, για να δούμε και να εξετάσουμε το τι έγινε. Και θα τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη μα και στη συζήτηση που θα γίνει. Και τα δικά σας σχόλια. Ευχαριστώ. Dziękuję bardzo. A na koniec sprawozdawca pan θα ακούσουμε τον ε, εισηγητή για τα τελικά σχόλια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλου του συναδέλφου που πήραν το λόγο. Ναι, παρατηρήσεις, πολύ ενδιαφέρουσε και πολύ σημαντικές. Θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω όσο μπορώ περισσότερο τα σχόλιά σας και θα συντάξω το νέο κείμενο. Θέλω να περιοριστώ σε κάποιες παρατηρήσεις, σε κάποιους προβληματισμούς από αυτούς που άκουσα. Η ιδέα του περιορισμού του χρόνου μεταφοράς αφορά μόνο τα ζώα προσφαγή. Είτε 8 είναι οι ώρες, είτε άλλο νούμερο, αφορά μόνο αυτά τα ζώα. Το νούμερο θα το συζητήσουμε. Ούτω ή άλλω δεν χρειάζεται το νούμερο να είναι το ίδιο για όλα τα είδη ζώων. Μπορούμε να αλλάξουμε ανά είδο ζώων. Σε ό,τι αφορά τα ζώα που μεταφέρονται για άλλου σκοπού, παραδείγματο χάρη τα υποειδή για του υπηκού αγώνε κτλ. Μην ξεχνάτε ότι και οι ίδιοι οδηγοί θέλουν να εξασφαλίσουν τις καλές συνθήκες μεταφοράς αυτών των ζώων. Ενώ ε, τα ζώα προσφαγή θεωρούνται ως προϊόν, ε, γιατί το, τα ζώα αυτά θα γίνουν κρέας. Ίσως να μην τους ενδιαφέρει λοιπόν τόσο πολύ η εξασφάλιση καλών συνθήκων μεταφοράς. Ε, αυτή η έκθεση λοιπόν αφορά αυτά τα ζώα, τα ζώα που μεταφέρονται προσφαγή. Λοιπόν, εγώ ως εισηγητής δεν ασχολούμαι μόνο με θέματα ευημερία των ζώων. Αν και προφανώς η ευμερία είναι πολύ σημαντική και είναι το πρώτο επίπεδο που θα εξετάσουμε. Αλλά ίσως να αρκεί κάποια στάση, ας πούμε, στον αυτοκινητόδρομο, εκεί στα, στους χώρους που παρκάρουν τα φορτηγά. Ε, μία μικρή στάση, ας πούμε, αρκεί για να ξεκουράσει τα ζώα, ίσως. Αλλά σε ορισμένε περιπτώσει ξέρουμε ότι υπάρχει κακή μεταχείριση των ζώων. Μερικές φορές το θέμα είναι πολιτιστικό, το θέμα είναι καθαρά πόσο πολιτισμένοι είμαστε. Ακόμα και από αυτή την πλευρά θα εξετάσω το θέμα του επίπεδου του πολιτισμού μας. Συχνά υπάρχει και το θέμα το οικονομικό. Ε, θα προσπαθήσω λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία να τα λάβω υπόψη μου και να τα εξισορροπήσω μεταξύ τους. Αν μεταφέρονται πολλά ζώα, ας πούμε, από την Πολωνία στην Ιταλία για να, να σφαγούν. Κάτι δεν πάει καλά στην αγορά. Και σίγουρα ποιος κερδίζει από αυτή τη μαζική μεταφορά ζώων, οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρηματίες που δημιουργούν αυτές τις εταιρείες μεταφοράς των ζώων, αυτοί κερδίζουν από αυτήν την ιστορία. Εμείς θα πρέπει να δούμε το θέμα πιο πλατιά δεν θα πρέπει να δούμε μόνο τα οικονομικά συμφέροντα των επιχειρηματιών, αλλά θα πρέπει να δούμε και τα ε, κοινωνικά θέματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών. Για τους καταναλωτές. Δεν θα ήταν καλύτερο να αγοράσουν ζώα, ας πούμε, Ιταλοί, Φερρυπίν, για να πάω το παράδειγμα που έθετα πριν, ε, που χρησιμοποιούσα πριν. Καλύτερο θα ήταν να αγοράζαν ζώα τα οποία είχαν εκτραφεί στην Ιταλία, παρά να αγοράζουν ζώα που μεταφέρονται από την Πολωνία. Γιατί τότε, ας πούμε, και όλες οι επιχειρήσεις στην Ιταλία θα είχαν περισσότερη δουλειά. Γιατί αν μεταφέρονται όλα τα, τα ζώα που εκτρέφονται στην Πολωνία, στην Ιταλία, Φερρυπίν, τότε οι Πολωνοί καταναλωτέ θα έχουν να αγοράσουν πολωνικό κρέα. Το οικονομικό συμφέρον, τα οικονομικά συμφέροντα, τα οικονομικά θέματα είναι προφανή. Ίσως ε, στο πρώτο σχέδιο του κειμένου μου τα οικονομικά θέματα δεν προέκυπταν τόσο σαφώς. Σας ευχαριστώ όλους εσάς που είπατε ότι πρέπει να επανέλθουμε στη λογική των μικρών τοπικών σφαγίων. Σωστό. Ούτως ή άλλως έτσι δημιουργούμε και μια οικονομική δραστηριότητα σε τοπικό επίπεδο και μειώνουμε και τις μεταφορές με όλο το κόστος και τις συνέπειες που υπάρχουν. Θα προσπαθήσω λοιπόν στο επόμενο κείμενο που θα ετοιμάσω να τονίσω περισσότερο, να προτάξω περισσότερο αυτά τα θέματα των μικρών σφαγίων. Ίσως ένα άλλο θέμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι το εξή. Γιατί κάτι λείπει στο κείμενό μου. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα χρηματοδότησης των μικρών εταιριών μεταποίησης που, έτσι, τις τοπικές επιχειρήσεις, ούτως ώστε ε, να γίνεται η σφαγή στον πλησιέστερο δυνατό τόπο ε, σε σχέση με τον τόπο εκτροφής. Αυτό είναι ένας άλλος τρόπος για να, μεταφέρ, να μειώσουμε τις ε, μεταφορές των ζώων από τη μια περιοχή στην άλλη. Υπάρχουν και γεωγραφικές διαφορές. Το συνειδητοποιώ τώρα αυτό. Κάτι που είναι δυνατό στο κέντρο της Ευρώπης, ο περιορισμός σε 8 ώρες Φερρυπίν, δεν είναι δυνατός σε άλλες περιοχές που δεν είναι στο κέντρο της Ευρώπης. Μπορεί, ας πούμε, οι 8 ώρες μπορεί να μην είναι δυνατές για τη Σουηδία, τη Φιλανδία ή την Ισπανία. Πρέπει τα ζώα να μεταφερθούν περισσότερες ώρες. οι αποστάσεις και οι γεωγραφικές διαφορές δεν μας επιτρέπουν να επιβάλλουμε τις 8 ώρες παντού. Τέλος πάντων, οι 8 ώρες θα μπορούσαν να είναι ένα σημείο αναφοράς, κατά την άποψή μου. Ο στόχος είναι να περιορίσουμε και κατ' να επιτρέψουμε τη μεταφορά για περισσότερο από 8 ώρες. την εξαίρεση την δίνουμε, ας πούμε, για γεωγραφικούς λόγους. Να, ένας λόγος. Ούτως ή άλλως, σε σχέση με το παρελθόν, οι συνθήκε μεταφορά και αυτό το λέει το κείμενο, έχουν βελτιωθεί. Αυτά, μάλιστα. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά θέματα που ακούστηκαν. Και με αυτά τα στοιχεία θα προσπαθήσω να εμπλουτίσω περαιτέρω το κείμενό μου θα εστιαστώ περισσότερο στο νέο κείμενο ε, στα μικρά σφαγεία. Αυτά, σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά όλους όσους πήρατε το λόγο. Α, ξέχασα και κάτι, το θέμα των ελέγχων. Για δεύτερη φορά εκλέγομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την πρώτη μου εκλογή ασχολήθηκα πάντα με αυτό το θέμα, με την ευμερία των ζώων. Και έχω κουραστεί να βλέπω ότι εγκρίνουμε και ψηφίζουμε κανόνες που επειδή δεν εφαρμόζονται ή επειδή είναι δύσκολο να εφαρμοστούν, τελικά γίνονται φαρσοκομωδία. Φέρει πίν. Ε, στην Ευρώπη έχουμε, δίνουμε τεράστια σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο, η κάθε χώρα έχει τον δικό της δημοσιολαβητή. Υπάρχουν διαφορετικές νομοθετικές διατάξεις σε κάθε χώρα. Αλλά, εν πάση έχουμε ένα καλό σύστημα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και, τέλος πάντων, όλες αυτές οι νομοθεσίες έχουν νόημα. Όλοι οι κανόνες, όμως, που αφορούν την ευημερία των ζώων, είναι απλώς λόγια, λόγια, λόγια του αέρα εφαρμόζονται ελάχιστα οι κανόνες και αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ. Α σκεφτώ την κατάσταση στη χώρα μου, την Πολωνία, όπου υπάρχουν οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ε, ζώων, υπάρχουν εθνικές διατάξεις, αλλά δεν υπάρχει κανένα φορέας εθνικός υπεύθυνο για ελέγχου. όλων αυτών των κανόνων. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η έλεγχοι. Παραδείγματο χάρη, υπάρχουν κτηνιατικοί έλεγχοι, κτηνιατρικέ ας που ασχολούνται με μια σειρά από θέματα. Αλλά την προστασία των ζώων είναι ένα από τα χιλιάδε θέματα που πρέπει να ελέγξουν. Επίση υπάρχουν και οι έλεγχοι στου δρόμου από την τροχέα. Και η τροχέα ας πούμε Α, αυτή μπορεί να ελέγξει ας πούμε, κάποια θέματα μεταφορά των ζώων. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι η προτεραιότητα τη τροχέα το να ελέγχει τη μεταφορά των ζώων. Καλό θα ήταν να έχουμε ένα φορέα λοιπόν που ασχολείται αποκλειστικά με θέματα προστασίας των ζώων. Σε μια χώρα όπως η Πολωνία, που είναι μεγάλη χώρα, ένας φορέας τέτοιος, με λίγα άτομα θα μπορούσε να εξασφαλίσει καλούς ελέγχους χωρίς ε, μεγάλο κόστος και έξοδα. Δεν νομίζω ότι για κανένα κρατός το κόστος θα ήταν μεγάλο από τη δημιουργία τέτοιων φορέων. αρχίζουμε να μιλάμε για την προστασία και την ευμερία των ζώων. Και όμω έχουμε τόσο διαφορετικά συστήματα στα διάφορα κράτη-μέλη. Σε ορισμένε περιπτώσει λειτουργούν καλά, σε άλλε περιπτώσει λειτουργούν άσχημα. Αλλά τελικά αφήνουμε, α πούμε, στον καθένα να κάνει ό,τι θέλει. Ίσως ευκαιρία είναι αυτή η έκθεση για να μας κάνει να σκεφτούμε και το ζήτημα των ελέγχων. Σε αυτή την έκθεση θα προσπαθήσω να μιλήσω για την ανάγκη δημιουργία ενός συστήματος πιο τακτικού, πιο οργανωμένου ε, που θα ελέγχει τα θέματα προστασία των ζώων. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα. Πρόεδρος, συμπεράσματα. Φτάσαμε στα συμπεράσματα. Θα ξανασχοληθούμε πολλές φορές ακόμα με αυτό το θέμα που είναι τόσο πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον. Μην ξεχνάμε όμως ότι δεν θα είναι εύκολο να ολοκληρώσουμε αυτή τη δουλειά, γιατί υπάρχουν διάφορα θέματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, διάφορα κριτήρια που πρέπει να σεβαστούμε κτλ. Με αυτά τελειώνουμε μια διήμερη πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση. Ε, σας θυμίζω στο όνομα του πρόεδρου μας, του κύριου Ντεκάστρο, ότι στις 19 θα γίνει μια συνεδρίαση για την ΚΑΠ. Και στις 19 λοιπόν του Μαρτίου θα κάνουμε και άλλες ενδιαφέρουσες συζητήσει. Μπορούμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη λειτουργία, τη λειτουργία της ε, γεωργικής πολιτικής. Αυτά ευχαριστώ.